Hello everybody who could make it. Apparently, you know, many of our colleagues, not apparently, but really, our many of our... Καλησπέρα σας. Πολλοί από τους συναδέλφους μας, από ό,τι φαίνεται, έχουν, ε, ε δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν λόγω των χιονοπτώσεων, των καταιγίδων κτλ. Θα ήθελα να σας πω κάτι που ήδη γνωρίζετε, ότι η ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Φαμπιός, που ήθελε να έρθει και να μας ενημερώσει, και να ακυρωθεί λόγω καιρικών συνθήκων και διακοπής των σιδηροδρομικών συνδέσεων ανάμεσα στις Βρυξέλλες και το Παρίσι. Αλλά αύριο το απόγευμα στις 3 η συζήτηση για τις δύο χρηματοδοτήσεις του κυρίου Σαλαφράγκα για την απαλλαγή 2011 αναβάλλεται και στη θέση της Στη θέση τους θα συζητήσουμε την κοινή ανακοίνωση της ΣΥΠΑ της και του Επίτροπου Φίλε για το Μαγρέμπ, Τη ε, την παρουσία του κυρίου Μιγκαρέλη, που είναι ο υπεύθυνο της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Έχουμε δε ε, προβλέψει συζήτηση για το Μαλί στη σημεία ανάμεσα στις 9.30 και τις 11.30 το πρωί ε, και για να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Νίκολας Βέσκοτ που είναι ο Γενικός Διευθυντής για την Αφρική και τον κύριο Walter Σίφενς που είναι ο Διευθυντής ε, για την διαχείριση κρίσεων και τον σχεδιασμό και οι δύο από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Και στις 23 ε, Ιανουαρίου μαζί με την ΤΕΒΕ θα συναντηθούμε για ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο της Σομαλίας Χασάν Σίκ Μαχμούτ. Στις 6 Φεβρουαρίου ανάμεσα στις 2 και 3 ε, το μεσημέρι. Η ΑΦΕΤ θα κάνει μια ανέκτακτη συνεδρίαση με τη Λουσίντα Κρέιτον, που είναι Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ιρλανδίας, για ενημέρωση για... σχετικά με το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ε, της 31ης Ιανουαρίου. Βλέπετε ότι πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά διαφόρων συνεδριάσεων που ξε... αρχίζουμε από τον Ιούλιο και φτάνουμε μέχρι και τον Οκτώβριο, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα θεωρήσουμε πως εγκρίνονται και θα περάσουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι η τροπολογία της... Η τροποποίηση, συγγνώμη, της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων. Ο κύριος Πάβελ Κόβαλ που είναι ο εισηγητής εγκρίνει την ε, συμφωνία αυτή όπως έχει τροποποιηθεί, αλλά επειδή απουσιάζει θα δώσω στον κύριο Τσάρλ Στάνοκ που είναι συντονιστή της ομάδας το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ζητώ συγγνώμη εξ του κυρίου Παύλ Κόβαλ ε, που λείπει και είμαι ευτυχής που εγώ είμαι εδώ παρά τις καθυστερήσεις του Eurostar και των κερικών συνθηκών της Βόρειας Γαλλίας. Βέβαια το θέμα αφορά την, ε, την ε, περιοχή Σέγγεν και άρα όχι τη χώρα μου. Απάντως η ομάδα, μας, ε, η ομάδα μου και εμείς στηρίζουμε αυτήν την τροποποίηση που είναι ένα μικρό βήμα προς την θέσπιση ενός καθεστώτος άνευ θεωρήσεων ανάμεσα στην Ουκρανία και την ΕΕ κάτι που η Ουκρανία έχει βγενός επιτρέψει για όλους τους πολίτες της Ένωσης, εντός και εκτός έγκεν, εδώ και δέκα χρόνια πια, ενώ εμείς διαπραγματευόμαστε ακόμα την πλήρη απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Εδώ πρόκειται για μια απλή διευκόλυνση με κάποιους περιορισμούς για όσους Ουκρανούς θέλουν να μεταβούν στην, στον χώρο Σέγγεν. Θα δείτε στη σελίδα 3 την σύντομη αιτιολόγηση. Δεν υπάρχουν τροπολογίες στη γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση βασικά στηρίζει την θέση της ΛΥΜΠΕ, δηλαδή να προχωρήσουμε και να εγκρίνουμε αυτήν την τροποποίηση που από ό,τι κατάλαβα χρειάζεται την νομοθετική φύση συμφωνία του Ευρωκοινοβουλίου, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που είναι δικές μας και αφορά πράγματα όπως η, παράταση, η επέκταση της κατηγορίας ανθρώπων που ζητούν βίζα για ε, ε, χώριση θεωρήσεων για ένα έως πέντε έτη για πολλαπλές εισόδους για τους ανθρώπους που που ταξιδεύουν στην Ένωση για εμπορικούς, ακαδημαϊκούς σκοπούς, για εκπροσώπους φοιτητών, για μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκπρόσωπους θρησκευτικών κοινοτήτων και ανθρώπους που συμμετέχουν σε διασκέψεις ή σεμινάρια που οργανώνονται στα επικράτεια της Ένωσης ή που χρειάζεται να μεταβαίνουν τακτικά στην Ένωση για ιατρικούς λόγους ή που καθώς και ε, σε, ε, μέλη της οικογένειας των ασθενών που μεταβαίνουν για ειδικέ αγωγέ τακτικά στην ε, επικράτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω λοιπόν, Πρόεδρε, πως όλα αυτά θα εγκριθούν χωρίς αντίρρηση από τα μέλη της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε δεν είναι εδώ για τους ίδιους λόγους που Λείπουν και άλλοι συνάδελφοι. Θέλω να παρουσιάσω τη θέση του ως στο ΕΛΚ. Ο κ. Προτασίεβης, ο σκιώδης εισηγητής, είναι και αντιπρόεδρος τη ομάδα υπεύθυνη για τις γειτονικέ χώρες και πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντική συμφωνία γιατί ενισχύει τις επαφές μεταξύ ανθρώπων. Ιδιαίτερα η διευκόλυνση των θεωρήσεων είναι σημαντικό εργαλείο γιατί προωθεί ευρωπαϊκές αξίες και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε ότι οι τροπολογίες είναι απαραίτητες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία μεταξύ, με την Ουκρανία γιατί απαλήφει κενά καταργεί επαχθείς διαδικασίες για φοιτητέ, εκπροσώπους ε, και μη κυβερνητικών οργανώσεων κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε ήταν υπέρ της κοινωνίας των πολιτών στις γειτονικέ χώρες. Οπότε αυτή η συμφωνία ευθυγραμμίζεται απόλυτα με αυτή την πολιτική, όπως και με την ενωσιακή πολιτική προς την, ε, τους εξανατολών γείτονες είναι απλή ψηφία και το ΕΛΚ θα ψηφίσει υπέρ. Ε, ευχαριστώ, κύριο Σίγκετς. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως δεν είναι αμφιλεγόμενη η συμφωνία αυτή, δεν παρουσιάζει προβλήματα. Αντικατοπτρίζει ένα πνεύμα συνεργασίας με την Ουκρανία και στη Σύνοδο Κορυφή ε, με, για την πολιτική γειτονία με του εξανατολών ε, γείτονε, ε, η Ουκρανία παρουσιάζεται ω χώρα υποδειγματική προκειμένου πέρι των διευκολύνσεων των θεωρήσεων. Όπως είπε πολύ σωστά και ο κύριο Στάνοκ, πρόκειται για μικρό βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω όμως ότι το βήμα αυτό θα το θα διαπιστώσουμε ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό αν ρωτήσουμε και το λαό της Ουκρανίας. Εμείς θεωρούμε στην Ευρώπη ότι είναι σημαντικό να πάρουν το σωστό μήνυμα οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις της Ουκρανίας. Δηλαδή ότι δεν εγκαταλείπει η Ευρωπαϊκή Ένωση την Ουκρανία, δεν απομακρύνεται από τη χώρα αυτή. μια διαδικασία ανολοκλήρωτη ακόμα είναι η διαδικασία για την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης. Αυτά που κάνουμε εμείς δηλαδή αποτελούν ε, σημαντικά μηνύματα για την Ουκρανία. Έτσι λοιπόν σημειώνουμε με ικανοποίηση την θέση σε ισχύ αυτής της συμφωνίας για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων Κάποιοι μάλιστα είπαν ότι λόγω λοιπόν μεταρρυθμίσεων θα έπρεπε να επιπλήξουμε την Ουκρανία. Έχω ακούσει και εγώ τέτοιες φωνές, αλλά νομίζω ότι δεν είναι σωστά τα επιχειρήματα αυτά. διότι εμείς θα πρέπει να προτάξουμε αυτά που είναι σημαντικά για τους πολίτες. Επίσης, έχουμε μελετήσει και κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά με την έκδοση των θεωρήσεων και παρατηρείται κάποια ανισορροπία, κάποιες ανισότητες γιατί κάποιες χώρες ακολουθούν πολύ περιοριστική πολιτική στην έκδοση των θεωρήσεων και περιμένουν σε μακριές ουρές οι ενδιαφερόμενοι και πολλές φορές τους αντιμετωπίζουν απαξιωτικά. Αυτή είναι μια κακή εμπειρία για τους ενδιαφερόμενους. Σε άλλες χώρες πάλι εκδίδονται εκατομμύρια θεωρήσεων και ενώ οι πρώτες χώρες μόνο κάποιες χιλιάδες μόνο. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σωστό το βήμα και μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και εγώ ευχαριστώ. Κυρία Νέιτ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, όπως και όλοι οι άλλοι, ακόμα και αυτοί που δεν ήρθαν λόγω καιρικών συνθήκων, θα ήθελα να πω εξ ονόματος λοιπόν της αντιπροσωπείας μου ότι εγκρίνουμε την πρόταση και θα την υποστηρίξουμε, θα την ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα για την Κομισιόν, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Δίτριχ Πάλμαν ή η Γκαμπριέλα Σμιτ. Θέλετε να παρέμβετε στο σημείο αυτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ και καλό απόγευμα. Είμαι ο Ντίτρεχ Μπάρμαν αναπληρωμα... Ε, αναπληρωτής διευθυντής ε, στην ε, διεύθυνση για τις θεωρήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ο συμφωνία για τον πληθυσμό γενικότερα στην Ουκρανία. Διευκολύνει πολλές κατηγορίες όπως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, νέους συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις, δημοσιογράφους και πολλούς άλλους που μπορεί να ωφεληθούν από τις πρόσθετες αυτές διευκολύνσεις. Θεωρούμε επίσης τη συμφωνία αυτή μια συμφωνία που πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, θα ήθελα να καταγραφεί ότι ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2008 η Συμφωνία για Διευκόλυνση των ε, Θεωρήσεων και εδώ ε, απλώς η Συμφωνία προσθέτει και άλλες διευκολύνσεις. Χαιρετίζω λοιπόν ε, την γνωμοδότηση του εισηγητού, παρόλο που ο ίδιος δεν παρευρίσκεται ε, σήμερα το απόγευμα και προσβλέπουμε σε γρήγορη ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα εντάξει και σε μετέπειτα στάδιο την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Ε, ο κύριος Κύριλοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι πρόσθετες διευκολύνσεις που θεωρώ ότι υποστηρίζονται από την πλειοψηφία των συναδέλφων είναι κάτι που σε εύθετο χρόνο, δηλαδή στο σωστό χρόνο στέλνει ένα μήνυμα κυρίως για τον λαό της Ουκρανίας, κυρίως τους νέους στη χώρα αυτή, τους φοιτητές Ε, και τι μη κυβερνητικέ οργανώσεις στην κοινωνία των πολιτών. Γιατί λέω ότι ε, στέλνετε το μήνυμα στο σωστό χρόνο. Βεβαίω ακόμα έχουμε πολλά προβλήματα να λύσουμε, ιδιαίτερα στην πολιτική της χώρας αυτής. Αλλά το μήνυμα είναι σωστό. Δίνει πρόσθετα κίνητρα στον Ουκρανικό λαό να παλέψει για τα δικαιώματά του, για μια καλύτερη κοινωνία, για την ανάπτυξη της χώρας ε, και προφανώς ε, και πάνω απ' όλα στέλνει το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση την χείρα ε, βοηθείας και θέλει να βοηθήσει τη διαδικασία της συνεργασίας και της περαιτέρω ολοκλήρωσης της Ουκρανίας και της ε, Ουκρανικής κοινωνίας. Το πολιτικό μήνυμα λοιπόν είναι σωστό και πρέπει όλοι να το υποστηρίξουμε. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Ανακοινώνω ότι η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο και δεν έχουν υποβληθεί τροπολογίες. Προχωρούμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα μας που είναι η έκθεση πρόοδου για το Μαυροβούνιο. Είναι η δεύτερη εξέταση του σχεδίου έκθεσης. Έχουμε 92 τροπολογίες και 8 συμβιβαστικές και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Τάνοκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όταν ε, παρουσίασα για πρώτη φορά αυτό το θέμα, μίλησα για πέντε λεπτά. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα ίδια και τώρα. Για να συνοψίσω πάντως, το Μαυροβούνι είναι μια καλή θετική ιστορία. Είναι μια μικρή και όμορφη χώρα. Δεν υποφέρει από τα μεγάλα προβλήματα που υποφέρουν κάποιες γείτονες προς αυτήν χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι λοιπόν μια συμπυκνωμένη χώρα με ελάχιστες ε, μικρής σημασίας διαμάχες. Η οικονομία μακροοικονομικά είναι σχετικά σταθερή, αν και παρόλο που χρησιμοποιούν το ευρώ, προσπαθούν ε, να τα βρούνε και με τους γείτονες. Είναι μια χώρα η οποία από τον Ιούνιο και μετά έχει το δικαίωμα να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις ως υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα. Η Σερβία είναι υποψήφια και βέβαια η Μακεδονία είναι μια χώρα που μπορεί να προχωρήσει εξαιτία τη διαμάχη τη με μία από τι χώρε μέλη μα. Το Μαυροβούνι λοιπόν πηγαίνει στην σωστή κατεύθυνση. Έχουν γίνει και κάποιες τροποποίησεις στην κυβέρνηση πρόσφατα, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές από την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Ο Πρωθυπουργό Λούξεν είναι πίσω. Ε, δεν είναι καν σαφές κατά πόσο έφυγε ποτέ από τον συνασπισμό επικεφαλής του κόμματός του και ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο κύριος Λούξη, είναι τώρα υπουργός εξωτερικών. Είναι μια έμπειρη ομάδα αυτή. Στο Λονδίνο πριν από δύο εβδομάδες μίλησα εκεί και συζήτησα και με τον πρέσβη του Μαυροβουνίου στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδερ Πέγιοβιτς. Είναι έμπειρη όλη η ομάδα που βρίσκεται στα νέα της χώρας αυτή τη στιγμή για να προχωρήσουν και στη δικαστική ε, εξουσία και για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλα τα θέματα, εν πάση περιπτώσει, που απασχολούν τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ, που είναι το οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά, η διαφάνεια, ε, δικαστική εξουσία κλπ. κλπ. Δικαιώματα μειονοτήτων. Η δικιά μου λοιπόν η έκθεση, που είναι σχετικά σύντομη, ε, πήρε 92 τροπολογίες, όπως είπατε κι εσείς. Υπάρχουν 8 συμβιβαστικές πάντως, όπου καταλήξαμε με τους κοιόδης συζητητέ στο Στρασβούργο και υπάρχει ευρεία συμφωνία πάνω σε αυτές με μια-δυο εξαιρέσεις. Η πρώτη απλώς ε, λέει ότι καλωσορίζει την απόφαση κτλ. Η κυρία Κόπα από τους σοσιαλιστές από ό,τι κατάλαβα θέλει να προσθέσει και ένα μέρος της τροπολογίας της 10 ως προφορική τροποποίηση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ από αυτού. Η συμβαστική 2 τώρα αναφέρεται στην εκλογική διαδικασία και το δικαίωμα ψήφου τη χρηματοδότηση των κομμάτων, τη διαφάνεια κλπ. Η συμβαστική 3 αναφέρεται πάλι στη δικαιοσύνη και άλλα θέματα όπως είναι τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων εφόσον κρατούνται βάσει του δικαστικού συστήματος. Υπάρχει συμβαστική 4 που αναφέρεται σε διάφορα κεφάλαια και εδώ έχει να κάνει με τη διαφθορά των θεσμών και ζητάει περισσότερη διαφάνεια στην χρηματοδότηση των κομμάτων, στην προεκλογική εκστρατεία κλπ. Η συμβαστική 5 μιλάει για την ελευθερία έκφρασης και τα μέσα ενημέρωσης. Κατά το παρελθόν υπήρξαν υπόνοιες για όχληση των ε, μέσων ενημέρωσης, για περιορισμό της ελεύθερης έκφρασης ε, έγιναν υπόνοιες για επιθέσεις κατά του τύπου. Υπάρχουν τέτοιοι ισχυρισμοί και λέμε ότι πρέπει να υπάρξει πρόοδος και εδώ ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει μια κοινωνία με διαφάνεια και με ελευθερία έκφρασης του τύπου και της τηλεόρασης. Είπαμε, είναι μια μικρή χώρα, οπότε είναι δύσκολο να υπάρχει απόλυτη ανεξαρτησία όπως έχουμε αλλού, αλλά εν πάση περιπτώσει αν μη τι άλλο οι εκδότες να είναι ανεξάρτητοι. Αυτά λέει η Συμβαστική 5. Συμβαστική 6 τώρα. Εδώ αναφερόμαστε στα δικαιώματα των μειονοτήτων. Υπάρχουν κάποιες από τους Ρώμα, τους Ασκάλι και την Αιγυπτιακή κοινότητα Κάποιοι από αυτούς έρχονται από το κοσυφοπέδιο και κάποιοι είναι σε καταβλισμούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λυθεί. Υπάρχει επίσης το θέμα των δικαιωμάτων των LGBT, ομοφιλόφιλοι κλπ. Στο Στρασβούργο είχαμε μιλήσει με κάποιους και σίγουρα πρέπει να φροντίσει η χώρα να ενισχύσει τα δικαιώματά τους, να μην υπάρχουν προβλήματα με την κατηγορία αυτή των πολιτών. Η Συμβαστική 7 αναφέρεται στα δικαιώματα των διοθήλων, των γυναικών ιδιαίτερα και την εκπροσώπηση των γυναικών στα δημόσια αξιώματα. Υπάρχουν και κάποια σχόλια για μακροοικονομικές στατιστικές, ε, για τα θέματα του πληθωρισμού, του χρέους και το γεγονός ότι είναι μια μικρή οικονομία που βασίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό στον τουρισμό. Δεν είναι αρκετά διαφοροποιημένη. Και πρέπει να γίνουν περισσότερα για να αντιμετωπιστεί η ανεργία και να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λέμε επίσης ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια σε διάφορες ε, περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με την κοινωνία. Γενικά πάντως πρέπει να σας πω ότι είναι τιμή για μένα που ασχολούμαι με την χώρα αυτή, μια χώρα ιδιαίτερα σταθερή και που ξεκάθαρα πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα έπρεπε να κρυθεί βάση των επιτευγμάτων της και δεν θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη προβλήματα που έχουν άλλες γείτονες προς αυτήν χώρες. Αυτά έχω να πω προς το παρόν. Και από εκεί και πέρα περιμένω τα σχόλια των συναδέρφων πάνω στις συμβαστικές κυρίως τροπολογίες, ώστε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα το προνόμιο να δουλέψω εδώ και κάποια χρόνια με τον Τσάρλ Στάνο και το Μαυροβούνιο και ήμουν ικανοποιημένη και από το πρώτο κείμενο που παρουσίασε γιατί το βρήκα ισορροπημένο. Και αντικατοπτρίζει η κατάσταση με ρεαλισμό. Βρίσκω όμως ότι το κείμενο με τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες θα είναι ακόμα πιο ισορροπημένο και βελτιωμένο. Υποστηρίζουμε όλες τις συμβιβαστικές τροπολογίες όπως και ένα μεγάλο αριθμό από τις ε, τροπολογίες, τις υπόλοιπε. Επίσης ξέρω ότι η κυρία Κοπά θα υποβάλει αύριο προφορική τροπολογία στην πρώτη συμβιβαστική και αυτή την προφορική τροπολογία εγώ επίση θα υποστηρίξω. Στο τέλος λοιπόν νομίζω ότι θα έχουμε ένα καλό και ρεαλιστικό κείμενο χωρίς να προβλέπω μεγάλα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκόμες. Ο σκιώδης μας δεν είναι εδώ, λόγω του χιονιού και εκείνος. Πρέπει να πω όμως, εξ ονόματός του, ότι εκφράζουμε ευγνωμοσύνη στον κύριο Τάνοκ για την καλή δουλειά και την καλή συνεργασία με όλους τους σκιώδεις. Και επιβεβαιώνω ότι δεν ε, έχουμε πρόβλημα και χαιρόμεθα διότι θα γίνει δεκτή η τροπολογία της κυρίας Κοπά Πόλους. Ο κύριος ε, Τάνοκ μίλησε λεπτομερώς για τα βασικά ε, προβλήματα, αν θέλετε, τις ανησυχίες που εκφράζουμε μέσα από τις 8 συμβιβαστικέ τροπολογίες. Πρέπει να πω ότι η περίοδος των διαπραγματεύσεων είναι κρίσιμη περίοδος για ε, μια αλλαγή στη χώρα. Είναι η περίοδος κατά την οποία θα ασκήσει μεγάλη επιρροή η Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουν οι αλλαγές, το ξέρουμε και από τις δικές μας χώρες. Μάλιστα ε, είδαμε ότι όταν προσχωρήσει κανείς υπάρχουν πολλά θέματα που πια δεν τίθενται, ερωτήσεις που δεν γίνονται και μάλιστα η χώρα μου είναι ένα καλό παράδειγμα όπου βλέπουμε να σημειώνεται σήμερα μια οπισθοχώρηση ακόμα και αν είχαμε προσχωρήσει χρόνια πριν. Σίγουρα ισχύει αυτό για τη χώρα μου όπου κάποια πράγματα που θεωρούσαμε ότι είναι κεκτημένο, ε, ευρωπαϊκό, τώρα οπισθοδρομούν λόγω των ε, τιμωρητικών πολιτικών συνταγών που επιβάλλονται. Ξαναγυρίζω στο Μαυροβούνιο. Είναι πολύ κρίσιμη αυτή η περίοδος λοιπόν κατά την οποία αλληλεπιδρά η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αρχές του Μαυροβουνίου και τις ε, για την κοινωνία των πολιτών για να υπάρξει αλλαγή. Γι' αυτό είναι κρίσιμη περίοδος. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών, ζωτικό θέμα, όπως επίσης και η καταπολέμηση της διαφθοράς, ε, η μάχη υπέρ της διαφάνειας του κράτους δικαίου, που επηρεάζουν όλα αυτά τόσο πολύ όλους τους άλλους τομείς. Αυτό το υπογράμμισε και ο κύριος Στάνοκ. Ε, θα πρέπει σε κεντρικό επίπεδο να ασχοληθούμε με αυτά γιατί λογοδοσία, διαφάνεια ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κεντρικό επίπεδο και εδώ κεντρικό είναι ο ρόλος των ε, μέσων ενημέρωσης που πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Εμείς μετά την ψήφιση της έκθεσης θα χρησιμοποιήσουμε την έκθεση για να ε, προωθηθεί η αλλαγή στο Μαυροβούνιο βεβαίως ε, πάντοτε μέσα από την κοινωνία και την κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ. Ο Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφος ε, που είναι σκιώδης για την ομάδα μου δεν ε, είναι εδώ, απουσιάζει, οπότε θα ε, παρέμβω εξ ονόματός του για λαγοριασμό του Άλντε. Καταρχήν, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή κύριο Τάνοκ για την έκθεση που συνέταξε για το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο είναι ένας από τους πρωτοπόρους στα Βαλκάνια και αποτελεί πρότυπο για όλες τις κοντινές του χώρες που είναι πολύ μεγαλύτερες. Ε, από τη μια πλευρά έχουμε τη Βοσνία Ερζεγοβίνη που δεν ξέρουμε τι θα κάνει ακολουθεί τη ρητορική του εθνικισμού και των συγκρούσεων, ενώ από την άλλη έχουμε το Μαυροβούνιο, το οποίο αναπτύσσει καλές ε, σχέσεις γειτονίας και δεσμεύεται για να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται προετοιμασία δε για τις προεδρικές εκλογές και αυτό θα είναι ένα πολύ κεντρικό βήμα, βασικό βήμα για τη χώρα. Ο Σέρβος Πρόεδρος μετέβει για επίσημη επίσκεψη στο Μαυροβούνιο. Ο κύριος Νίκολιτς. Ξέρετε ότι δεν μπορεί ας πούμε, να πάει στην Κροατία λόγω κάποιων επίμαχων δηλώσεων ε, στο παρελθόν. Μπορεί λοιπόν η πρόσκληση αυτή να είναι ένας καλός ιονός για τα ε, Δυτικά Βαλκάνια. Εύχομαι ότι αργά ή γρήγορα θα μπορέσει να υπάρξει μια επαφή ανάμεσα στον Νίκολιτς και τον ε, πρόεδρο του Κωσυφοπεδίου πράγμα το οποίο ήδη είχε προβλεφθεί στο Μαυροβούνιο, αλλά δεν υλοποιήθηκε. Θα ελπίσουμε όμως ότι θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για μια τέτοια συνάντηση. Επίσης ε, πρέπει να συγχαρούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που άνοιξε στη συζήτηση τα πιο δύσκολα κεφάλαια, το 23 δηλαδή και το 24. Και όταν μετά θα δούμε και την έκθεση για την Τουρκία και για αυτό το θέμα και για την Τουρκία, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση για τα 23 και 24, όπου γίνεται λόγος για κράτος δικαίου, για ανθρώπινα δικαιώματα και για τα πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο και τη διαφθοράς. Θα πρέπει λοιπόν να επενέσουμε το Μαυροβούνιο γιατί αν ξεκίνησε και έκλεισε τη συζήτηση για το κεφάλαιο για τις επιστήμες και την έρευνα. Πράγμα που αποδεικνύει ότι το 2013 το Μαυροβούνιο θα είναι σε θέση να ξεκινήσει τη καινούρια κεφάλαια. Ο Τάνοκ, ο κύριος Τάνοκ ε, εξάλλου προσφέρει αποδεκτές λύσεις τόσο για τους ομοφιλόφιλους, λεσβίες και τα λοιπά, όσο για τους άνδρες και τις γυναίκες και εξ ονόματος της Άλντε λοιπόν. Εμείς στηρίζουμε τη συμβιβαστική τροπολογία και θα την υπερψηφίσουμε. Και επίσης ε, να πω ότι ο Υπουργό που ορίστηκε από το Μαυροβούνιο για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση είναι ένα άνθρωπο ο οποίος θα βοηθήσει τη χώρα του στο μονοπάτι προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Τάνοκ και είμαι βέβαιο ότι με αυτή την έκθεση θα καταφέρουμε να ενθαρρύνουμε τη χώρα αυτή να επιταχύνει την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι θα βοηθήσει και τις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων δείχνοντας πως ε, η διεύρυνση είναι ζωντανή και πολύ σημαντική για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, ότι ανάγνωση και συζήτηση της έκθεσης είχαμε την ευκαιρία, είχα την ευκαιρία ως κοιόδης εκ μέρους της ΓΚΟΕ να πω τις θέσεις μας σχετικά με τα θέματα της διεύρυνσης και ειδικά της ενταξιακής προοπτικής στο Βαλκανίο. Ε, συμφωνώ με τον εισηγητή μας ότι το Μαυροβούνιο μοιάζει να είναι από τις πιο εύκολες περιπτώσεις έναντι των άλλων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε απαιτητικοί όσο αφορά την έκθεσή μας. Ο στην έκθεση του εισηγητή υπάρχουν πράγματα με τα οποία συμφωνούμε, υπάρχουν πράγματα με τα οποία διαφωνούμε και υπάρχουν και ελλείψεις που νομίζουμε ότι χρειάζονταν να μπουν. Για το τελευταίο, καταθέσαμε σχετικές τροπολογίες. Ο εισηγητής δεν συμφωνεί με αυτές, θα τις αναφέρω, είναι τρεις. Παρά τα αυτά, παρακολουθώντας τη διαμόρφωση της έκθεσης, θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε και στον εισηγητή μας, ότι σε σχέση με τις οχτώ συμβιβαστικές προτάσεις, εμείς συμφωνούμε με την πρώτη πρόταση για την πρόοδο που έχει γίνει, συμβιβαστική τροπολογία, με την τρίτη για τα θέματα δικαιοσύνης, με την πέμπτη όσο αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την έκτη όσο αφορά τα δικαιώματα και την έβδομη η αναφορά για τις γυναίκες. Με αυτές τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες, παρότι δεν περιλαμβάνουν δικές μας νήξεις, ε, συμφωνούμε. Θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι προφανώς δεν συμφωνεί ο συγητής μας, αλλά υπάρχει περιπτώσει εγώ θέλω να το πω, εκεί που καταθέσαμε τις τροπολογίες, είναι τρία σημεία. Το ένα ότι απουσιάζει σοβαρή αναφορά στα δικαιώματα των εργαζομένων, στο θέμα της μείωσης της ανεργίας και στην δημιουργία δικτύου κοινωνικής προστασίας των φτωχών και των ανέργων. Διαβάζοντας όλες τις τροπολογίες, νομίζω ότι η κυρία Λούνατσεκ και η κυρία Κορνέλιασον έχουν κάνει τις ίδιες τροπολογίες. Θα τις υποστηρίξουμε στην ψηφοφορία. Η δεύτερη κατηγορία είναι για τροπολογίες που τονίζουμε ότι χρειάζονται δημόσιες επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού στην παράκτια τουριστική ζώνη. Και εδώ από την πλευρά της κυρίας Λούνατσεκ έχει κατατεθεί ε, τροπολογία που ζητάει ρήτρα σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη, ρήτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Και τέλος, ε, καταθέσαμε τροπολογία, δεν γίνεται δεκτή, ε, νομίζουμε ότι θα χρειαζόταν, στον τομέα της διαφθοράς και γενικά της υψηλής διαφθοράς, υπάρχουν θέματα που έχουν σχέση με τις ιδιωτικοποίησεις και τις ξένες επενδύσεις, που ελέγχονται για διαφθορά και θα το έλεγα με μια έκφραση διαφθορά εκτεταμένη όσον αφορά τα συμφέροντα της χώρας. Αυτές, αυτά είναι σημεία που καταθέσαμε συμπληρωματικές τροπολογίες. Αυτή είναι η δική μας ε, άποψη. Την τελική μας θέση θα την καθορίσουμε αύριο κατά την ψηφοφορία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Λούνατσεκ. Είσαστε έτοιμοι τώρα. Να παρέμβετε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Και συγγνώμη που καθυστέρησα. Δεν περίμενα ότι θα είχατε προχωρήσει τόσο γρήγορα με την Ουκρανία. Γι' αυτό. Δεν άκουσα βέβαια την παρουσίαση του κύριου Τάνοκ, αλλά τα συζητήσαμε, οι σκιώδεις συζητητές, και τον ευχαριστώ πολύ για την καλή δουλειά που έχει κάνει. Έχει ετοιμάσει μια καλή έκθεση, η οποία αναφέρεται σε όλα τα προβλήματα, ή τέλο πάντων σε όποια προβλήματα προέκυψαν. Το αναγνωρίζουμε αυτό. Και η ομάδα μου τον ευχαριστεί επίσης επειδή συζητάει την προσχώρηση αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Μαυροβούνιο. Είναι πάρα πολύ καλό γιατί είχαμε την Κροατία και είναι πολύ σημαντικό τώρα να έχουμε μια άλλη χώρα η οποία μπαίνει στο αυλάκι και εκείνη για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να ακολουθήσουν κι άλλες φέτος. Υπάρχουν τώρα τρεις πτυχές τις οποίες θα ήθελα να αναφερθώ από πλευράς των πρασίνων. Έχουμε κάποιες τροπολογίες που δεν είναι στις συμβαστικές, αλλά που θα θέλαμε να ζητήσουμε από τους ευρωβουλευτές να τις υπερψηφίσουν αύριο. Η μία έχει να κάνει με το θέμα των ομοφιλόφιλων και λοιπά στο Μαυροβούνιο. Θέλω να το πω και να επιμείνω ότι στις συμβαστικές και στο κείμενο σε σύγκριση με το τι γίνεται σε άλλες χώρες, υπάρχει πρόοδος στο Μαυροβούνιο. Έχουν ε, αναλάβει κάποια θετικά βήματα εκεί. Υπήρξε μάλιστα και μία διάσκεψη με υπουργούς για το θέμα της μη διάκρισης σε βάρος των ε, ΛΟΑΕΒ. Υπάρχει λοιπόν κάτι που θέλουμε οι κυβερνήσεις να το στηρίξουν, να μπορεί να γίνει φέτος αυτή η πορεία που γίνεται παραδοσιακά, η περίφημη parade, και γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να το υπερψηφίσετε αύριο. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα όμως που υπάρχει πολύ στο κείμενο που είναι η διαφθορά. Η διαφθορά ακόμα είναι πρόβλημα στο Μαυροβούνι. Και έτσι είναι καλό Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει, έχει αρχίσει, ίσως με τα κεφάλαια 23 και 24 στην διαδικασία διαπραγματεύσεων. Υπάρχει και μια πρόσφατη εξέλιξη που εμείς με την τροπολογία μας θέλουμε να καλύψουμε και αυτή είναι ότι η αδερφή του κ. Τζουκάνεβιτς ξεκίνησε νομική διαδικασία σε βάρος δύο δημοσιογράφων από δύο διαφορετικές εφημερίδες οι οποίοι έγραψαν για το άτομό της ε, αφήνοντας υπόνοιες ότι είχε προχωρήσει σε κάποιες παραβατικές συμπεριφορές. Νομίζω ότι και αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στην έκθεση και ζητάω την στήριξή σας. Και έρχομαι και στο τελευταίο που είναι η τροπολογία 82, η οποία ζητάει από τις αρχές να έχουν μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στις οικονομικές ε, εξελίξεις και την περιβαλλοντική προστασία. Ξέρετε ότι στο Σύνταγμα του Μαυροβονίου γίνεται μνήα για το ότι πρόκειται για μια οικολογική χώρα. Πρέπει λοιπόν να γίνουν περισσότερα, πιστεύω, να αναφέρουμε τον τουρισμό, γιατί η χώρα θέλει να προσφέρει καθαρό περιβάλλον στον τουρισμό και θέλει επίσης και ανάπτυξη στις ακτές κυρίως όπου όμως κινδυνεύουν από υπερβολική ανάπτυξη, γιατί αυτό θα είναι σε βάρος της περιβαλλοντικής προστασίας. Είναι πολύ ωραίο να θέλει κανείς να πάει να δει το ωραίο τοπία, την καθαρή θάλασσα. Συνεπώς εδώ δεν χρειαζόμαστε μόνο μέτρα κατά της ρήπανσης και υπέρ του περιβάλλοντος, αλλά χρειάζεται να δουλέψουμε επίσης και προς την κατεύθυνση της καλύτερης ανάπτυξης, ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο οικολογικός χαρακτήρας αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον κύριο Τάνοκ για το έργο του και για την καλή συνεργασία που είχαμε όλοι μαζί, οι σκιώδες μαζί του. Ελπίζω τις δικές μας τροπολογίες των Πρασίνων οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές να τις στηρίξουν αύριο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριε Κοπά τώρα. Thank you very much. Uh, I would like also to congratulate uh, the... Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή καταρχήν για την έκθεσή του που εντοπίζει τα βασικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία ε, ολοκλήρωσης του Μαυροβουνίου. Το Μαυροβουνίο έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χάρη στη συνένεση που έχει βρεθεί με, ανάμεσα στα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα και τις εθνοτικές ε, κοινότητες ε, σε σχέση με την ανάγκη να ληφθεί σοβαρά υπόψη η διαδικασία ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει αυτό να είναι σαφώ μήνυμα προ την γειτονική Αλβανία και Βοσνία Ριζογοβίνη, καθώ και να λειτουργήσει ω κίνητρο ώστε να ακολουθήσουν την ίδια πορεία. Είναι καλό να έχουμε υπόψη μα ότι το Μαυροβούνιο είναι η πρώτη χώρα όπου ε, εφαρμόζεται η νέα διαπραγματευτική προσέγγιση. Αυτό δεν είναι ευρέω κατανοητό και συχνά οδηγεί σε παρανοήσει. Ωστόσο πιστεύω πω μια ε, ε, νέα διατύπωση της, του εκτιμώντας ε θα ήταν καλή για να τονιστεί η σημασία του θέματος του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών θεμάτων. Επίσης θα πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες, να ενταθούν μάλλον οι προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου, η καταπολέμηση ε, του οργανωμένου εγκλήματος ε, και τη διαφθορά στα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων καθώς και η κατοίκων βία. Ευχαριστώ το τον κύριο Τάνοκ που δεν έχει παραμελήσει τα προσφυλή αυτά θέματα στο σχέδιό του και επειδή ανέπτυξε περαιτέρω την διατύπωση στη Συμβαστική 7. Όμω η Συμβαστική 7 δεν συμπεριλαμβάνει την τροπολογία υπαρθμών 60 που τονίζει ότι χάρη στην εισαγωγή των ποσοστώσεων περιφύλου στον εκλογικό νόμο οι γυναίκε για πρώτη φορά έχουν δυνατότητα να συμμετέχουν μαζικά στι εκλογέ. Μάλιστα, ένα σύνολο 264 γυναικών ήταν υποψήφιοι ψηφοψηφία τον περασμένο Οκτώβριο και ε, μια, ένα ψηφοδέλτιο είχε γυναίκα αρχηγό. Αυτή η βελτίωση αναγνωρίστηκε από τον ΟΑΣΕ και από τις ε, ε, οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών επί το Ελπίζω λοιπόν πω αυτή η τροπολογία 60 θα στηριχτεί κατά τη διάρκεια τη ψηφοφορία ω επιβεβαίωση μια πραγματική προθυμία να δούμε περισσότερε γυναίκε εκλεγμένε στο Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αγκουράκης. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε θα συνεχίσω στα ελληνικά. Να κερδίσουμε και χρόνο. Ε, καταρχήν, πριν, πριν να πω μερικές σκέψεις στην ε, έκθεση προόδου για την ένταξη του Μαυροβουνίου, ε, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σας εκφράσω την έντονη διαμαρτυρία μου για το γεγονός ότι ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας τελικά ανέβαλε το ταξίδι του και τη συζήτηση που είχαμε για τις πολύ σοβαρές και επικίνδυνες εξελίξεις στο Μαλί. Εγώ δεν πείθουμε για το επιχείρημα του, του καιρού. Νομίζω ότι είναι μια υποτίμηση ως προς την ε, Επιτροπή μας και αυτό λέει πολλά πράγματα. Τώρα, για την έκθεση όσον αφορά την ε, ενταξιακή διαδικασία για το Μαυροβούνιο. Όπως ε, θα ξέρετε και εσείς και οι συνάδελφοι, ε, το κόμμα μου τάσεται από άποψη αρχής ενάντια στη διεύνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί θεωρεί ότι η πολιτική που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα οξύνει ακόμα περισσότερο τα οξυμένα προβλήματα που έχουν οι χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη της. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, δεν θα σταθώ σε αυτό, θα σταθώ στην έκθεση. Ε, στην έκθεση ε, θα ήθελα να, να σημειώσω τέσσερα ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ενώ ό,τι γνωρίζουμε ότι η τωρινή καπιταλιστική κρίση και οι διαδικασίες της ένταξης, οι αναδιαρθρώσεις οι οποίες ζητούνται συνοδεύονται από ε, πολιτικές ιδιωτικοποιήσεων που έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο θέμα της απασχόλησης είτε για την πόλη μιλάμε είτε για το χωριό η έκθεση δεν κάνει καμία αναφορά στα ζητήματα αυτά. Φαίνεται σαν να απασχολεί το γεγονό ότι στη χώρα αυτή υπάρχουν ε, πάρα πολλοί άνεργοι και το τι θα γίνει με αυτού του ανθρώπου στο μέλλον. Δεύτερο ζήτημα δεν, δεν αφορά την έκθεση καθόλου τα ζητήματα των κοινωνικών υποδομών. Φυσικά γίνεται μια, μια αναφορά εκεί που γίνεται λόγος για τη μεγάλη φτώχεια, για τη μεγάλη φτώχεια των παιδιών και γίνεται μια αναφορά ότι αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, αλλά οι υποδομές δεν αφορούν μόνο θέμα παιδιών, αφορούν θέματα παιδείας, υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος, ενδεχομένως συγκοινωνιακά δίκτυα, δημόσιες μεταφορές, οι οποίες η έκθεση θεωρεί ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα ζητήματα αυτά και δεν αναφέρεται καθόλου. Τρίτο ζήτημα το οποίο το θεωρώ λάθος και απαράδεκτο είναι το σημείο 14 όπου η συγκητή συγχαίρει το Μαυροβούνιο για την διατήρηση της μακροοικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας, όμως δεν μας λέει ότι αυτή η μακροοικονομική και δημοσιονομική σταθερότητα έχει πάει τη χώρα πίσω. Δεν έχει λύσει τα προβλήματά της, αντίθετα έχει οξύνει και δεν φαίνεται να προτείνει και κάτι για το ζήτημα αυτό. Επίσης, ένα πέμπτο σοβαρό ζήτημα είναι αυτό που, στο οποίο γίνεται λόγος για την ε, ε, ε, για την συμμετοχή των ΜΚΟ στις ομάδες εργασίας που ασχολούνται με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Καταρχήν δεν, δεν διευκρινίζεται για ποιες ΜΚΟ γίνεται λόγος. ΜΚΟ υπάρχουν χιλιάδες στη χώρα αυτή, δεν ξέρουμε για ποιες μιλάμε. Δεύτερον, και το οποίο είναι ακόμα πιο σημαντικό, καλό θα είναι από τη στιγμή που χαιρετίζουμε αυτές τις συμμετοχές να έχουμε συνοπτικά για τις απόψεις των ΜΚΟ για τις διαδικασίες ένταξης, τις οποίες δεν τις έχουμε στην έκθεση και δεν τις έχουμε και σε αντίστοιχα ντοκουμέντα. Και τέλος το ζήτημα αυτό θα ήθελα να πω ότι πολύ πιο σημαντική είναι η τοποθέτηση των πολιτικών κομμάτων για τα οποία έκθεση τίποτα στις διαπραγματεύσεις για την ε, ε, ένταξη της χώρας. Ε, ένα τελευταίο ζήτημα είναι τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Σημειώνεται η ευχή των Μαυροβούνιων να επιλύσει τα ζητήματα με τα, ε, τα συνοριακά που υπάρχουν με τους γείτονές τους, αλλά δεν μας λέει τουλάχιστον σε ποια βάση θα είναι στη βάση του ΟΗΕ, θα είναι σε άλλη βάση, ποια βάση θα είναι αυτή. Και εμεί νομίζουμε ότι θα έπρεπε να είναι στη βάση του ΟΗΕ. Τέλο, κλείνω κύριε Πρόεδρε και σα ευχαριστώ για την υπομονή σα. Εγώ δεν συμφωνώ με την αναφορά στο σημείο 20 που γίνεται λόγο ε, να υιοθετήσει το Μαυροβούνιο την κοινή θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο ε, που έχει τόσο ολέθριο ρόλο παίξει ειδικά στην πρώην Ιουκοσταβία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Well, Σας ευχαριστώ. Η γενοδορία θα πρέπει να... Ε, και οι για αυτήν θα πρέπει να απευθυνθούν προς τον κύριο Λοράν Φαμπιού, γιατί αυτός ακύρωσε την επίσκεψη ε, και γι' αυτό έχουμε περισσότερο χρόνο, αλλά όπως είπαμε θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε την κατάσταση στο Μαλί με εκπροσώπους της γαλλικής κυβέρνησης. Τώρα, από την Κομισιόν έχουμε τον κύριο Λάγκε που αντιπροσωπεύει τη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνση. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ενημερώσω το Κοινοβούλιο για μια πρόσφατη επαφή του Πρόεδρου Μπαρόζο με τον Πρωθυπουργό Τσουκάνοβιτς που έγινε μάλιστα σήμερα το πρωί. Από ό,τι κατάλαβα, ήταν ένα από τα πρώτα ταξίδια του Πρωθυπουργού ε, Στι Βρυξέλλε ήρθε λοιπόν για να ευβεώσει την προσήλωσή του στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση για τον ίδιο και την κυβέρνησή του. Και επίσης μας ανέφερε την πρόοδο που σημειώνει το Μαυροβούνιο στην θέσπιση των δομών για να μπορέσουν να, να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει. Τώρα έχουν δημιουργηθεί 19 ομάδε εργασία και οι υπολοιπόμενε θα δημιουργηθούν πολύ σύντομα. Μιλάμε για τα κεφάλαια 23 και 24, τα κεφάλαια δηλαδή του κράτους δικαίου που αναφέρθηκαν ήδη εδώ ε, εργάζονται για, τα πρόγρα... για το σχέδιο εργασίας, πρόγραμμα εργασίας, προγράμματα δράσης με στόχο να υιοθετηθούν όλα αυτά την άνοιξη από την κυβέρνηση. Εν γέννη, καλωσόρισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμή στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Ξέρετε ότι είμαστε στα ε, μέσω μιας διαδικασίας screening, ελέγχου και αναμένεται πως ακόμα ένα κεφάλαιο θα ανοίξει υπό την Ιρλανδική Προεδρία. Ο πρόεδρος Μπαρόζο τόνισε την ανάγκη για την τροποποίηση του συντάγματος ώστε να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και νέα συστάσεις από την Αρμόδια Επιτροπή και επίσης ενθάρρυνε τον Πρωθυπουργό να έρθει σε επαφή με την Κροατία ώστε να βρεθεί λύση για την υπόθεση Βεφλάκα και να μπορέσει να προχωρήσει η κατάσταση. Το άλλο θέμα που πιστεύω ότι θα σας ενδιαφέρει είναι ότι την Παρασκευή ανακοινώθηκε η ημερομηνία για τις επόμενες προεδρικές εκλογές που θα γίνουν στις 7 Απριλίου με δεύτερο γύρο στις 15 Απριλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Θέλετε να κλείσετε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ιμπρισέζιτς. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία και Πραγματικά μου έχει δώσει πολλές συμβουλές γιατί είναι ειδικό στην περιοχή και καταλαβαίνει και τη γλώσσα και τον πολιτισμό των χωρών και με έχει βοηθήσει πολύ στη σύνταξη της έκθεσης. Ε, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκόμες για τα καλά της λόγια και την κυρία Κοπά που επίσης έδειξε το θέμα βέβαια ότι έχει υπάρξει ένα ε, αυστηρότερο όριο για είσοδο των χωρών μετά από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Όντω, οι χώρε αυτέ θα πρέπει να δουλέψουν πολύ περισσότερο από ό,τι πριν από 10 χρόνια, για παράδειγμα. Ε, και να ευχαριστήσω και τον κύριο Κατσίν που μίλησε εξ ονόματο τη Άλντε. Το Μαυροβούνιο είναι μόνο του, γιατί είναι η μόνη βαλκανική χώρα που είναι σε διαπραγματεύσει και έχουν και οι προεδρικές εκλογές που έρχονται και φυσικά αναφέρονται το γεγονός ότι ένα κεφάλαιο έχει, ήδη κλείσει αυτό που αφορά την έρευνα και την επιστήμες. Ήταν επιτυχής η επίσκεψη του Προέδρου της Σερβίας που ήταν εκεί, από ό,τι κατάλαβα, ήταν εκεί για την κηδεία ενός πρώην Υπουργού της Ιουκοσλαβίας. Δεν συμφωνώ όμω με τον κύριο Αγκουράκη, ίσως μην σας εκπλήσει αυτό, ε, ούτε με τον κύριο Χουντή της Γκουέ, γιατί ίσως να είναι ικανοποιημένοι που σε αυτή την περίπτωση δεν συμπεριέλαβα καθμία αναφορά ε, για συμμετοχή στο ΝΑΤΟ που την άλλη φορά του εξαγρίωσε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, δεν μπορώ να συμφωνήσω με τις απόψεις της Γκουε, ιδιαίτερα με τον κύριο Γκουράκη που είναι κατά διεύρυνση γιατί βλέπει μόνο την Ένωση ως μια λέσχη καπιταλιστών κατά τη ιδιωτικοποίηση κατά τη ευελιξίας των αγορών εργασίας. Εγώ ε, και να σας πω κύριε και να σας ενημερώσω κύριε Γκουράκη, η διαμάχη για τα σύνορα είναι με την Κροατία και είναι ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και αυτό θα πρέπει να επιταχυνθεί. Κάπως έχει κολλήσει, δεν έχει κινηθεί καθόλου το τελευταίο καιρό, αλλά αυτό είναι διμερές ζήτημα φυσικά. Τώρα, όσον αφορά την κυρία Λούνα Τσέκα και τις προβληματισμούς, ε, κάλυψα εκτεταμένα κυρία Λούνα Τσέκα το θέμα των δικαιωμάτων των ε, ε, ομοφιλόφιλων ε, και τα λοιπά όσον αφορά το θέμα της Pride, αυτά είναι θέματα εσωτερικής απόφασης, δεν είναι κατά της σχετικής παρέλασης, όχι από ό,τι κατάλαβα, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι κάνουν, πάντως βασική μου έμφαση δίνεται στην κατάργηση των διακρίσεων. Επίσης αναφέρατε ένα συγκεκριμένο θέμα μιας δικαστικής υποθέσεως που αφορά την αδελφή του, του Πρωθυπουργού. Κοιτάξτε να σας πω ότι εγώ σέβομαι την Βρετανική συν, ε, σύμβαση ότι δεν αναφέρουμε δικαστικές υποθέσεις που είναι υπό εκδίκαση μπορεί να, να διώξει ποινικά οποιαδήποτε εφημερίδα αν θεωρεί ότι έχει δυσφημιστεί. Ε, αν όντω ε, είναι λυπή στη δικασία και ε, αν υπάρξουν στοιχεία καταστολής της ελευθερίας του τύπου, τότε θα έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Αλλά σίγουρα εγώ δεν θέλω να υποστηρίξω τροπολογίες ώστε να γίνει δίκη πριν να έχει εξαντληθεί το ίδιο το δικαστικό το σύστημα, εφέσεις και λοιπά μέσα στο ίδιο το Μαυροβούνιο. Τώρα, οικονομική ανάπτυξη και περιβάλλον. Πολύ λεπτό θέμα, ούτε και δεν θέλω να υποδείξω λύσεις. Το Μαυροβούνι είναι ε, κυρίαρχη χώρα. Δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε για το ποια ακριβώς ισορροπία θα πρέπει να τηρήσουν. Έχουν το δικό τους κοινοβούλιο, δημοκρατικά εκλέγεται. Ε, ε, έχουμε πει πολλά για τη διατήρηση των περιβαλλοντικών στάνταρ και εκείνοι πρέπει να το αποδείξουν πλέον ότι το κάνουν στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν... Ε, γενικά, οι περισσότεροι σκιώδεις εισηγητές μίλησαν εξ ονόματος της ομάδας, στήριξαν την εκθεσή μου και τους ευχαριστώ γι' αυτό και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, όπως είπατε, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 9. Ακριβώς. Α, δεν έχει πέσει χιόνι βέβαια πάλι και δεν μπορούμε να φτάσουμε στο κοινοβούλιο. Αλλά πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο, έχουμε, που είναι η έκθεση πρόοδου για την Τουρκία, θα ήθελα να αναγνωρίσω και να σας ενημερώσω, να καλωσορίσω τα μέλη του Προεδρείου της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που είναι παρόντες εδώ. Και να σας πω ότι πρόκειται για την πρώτη εξέταση του σχεδίου ψηφίσματος για την ε, έκθεση πρόοδου της Κομισιόν για την Τουρκία για το 2012 και η κυρία Όμεν Ρόιτεν είναι εδώ μαζί μας. Θα τη δώσω το λόγο αμέσω και θα ήθελα να ανακοινώσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 5η Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Στις 12 το μεσημέρι που σας είπα, κυρία Όμεν Ρόιτεν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πέρυσι μιλήσαμε για την αλληλεξάρτηση που έχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία και πώς αυτή η αλληλεξάρτηση θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα στα πλαίσια μιας αμοιβαίας δέσμευσης. Τώρα, η εφαρμογή της θετικής ημερήσιας διάταξης το 2012 στα πλαίσια της αμοιβαίας αυτής δέσμευσης και σαφών στόχο. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι πράγματι η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να προχωρήσουν σε διάλογο, μπορούν να πετύχουν αμοιβαία κατανόηση και μπορούν επίσης να παράγουν θετικές αλλαγές. Όμως, τώρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα διατηρηθεί αυτή η επικοδομητική σχέση μέσα σε μια ατμόσφαιρα αμοιβαίας κατανόησης και αμοιβαίας και αμοιβαίου σεβασμού. Ειλικρινή πιστεύω ότι η ανανέωση των δεσμεύσεων στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγματεύσεων είναι κάτι που χρειάζεται. Για να καταλήξουμε σε αυτήν την ανανέωση της δέσμευσης χρειάζονται προσπάθειες εκατέρωθεν. Κύριε Πρόεδρε, η φετινή έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαστικής εξουσίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το πακέτο για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος αναφίβολα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, αλλά είναι πολύ βασικό να συνεχιστεί, να συνεχιστεί δηλαδή η μεταρρύθμιση των διαδικασιών και του πακέτου. Η κύρια προτεραιότητα επ' αυτού είναι να ασχοληθούμε με θέματα που έχουν να κάνουν με τους ευρύς ορισμούς που υπάρχουν όσον αφορά τα παραπτώματα και τις παραβιάσεις του ποινικού δικαίου αλλά και της τρομοκρατίας. Είναι πολύ βασικό να προωθήσουμε την ελευθερία της έκφρασης στην Τουρκία. Αγαπητοί συνάδελφοι, Πρόεδρε, η Τουρκία αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να προχωρήσει στις προσπάθειές της, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και εκείνη να κάνει ό,τι μπορεί για να τη βοηθήσει στη διαδικασία αυτή να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι που θα οδηγήσουν σε έναν ε, χάρτη πορείας για να δώσουμε νέα όθεση στη διαδικασία. Το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24, κατά τη γνώμη μου, θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Θέλω επίσης εδώ να υπογραμμίσω και το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, περιμένει και παρακολουθεί τις μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι ένας πολύ σημαντικός ε, στρατηγικός παίχτης και έχει πολύ μεγάλη σημασία για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, ο πολιτικός διάλογος πρέπει να ενισχυθεί και θέλω να ενθαρρύνω την Τουρκία να προχωρήσει στην πολιτική της υπέρ του διαλόγου σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως πάντα λέμε, η Τουρκία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και όσον αφορά τη Συρία. Γιατί έχει δεσμευτεί υπέρ των δημοκρατικών δυνάμεων στη Συρία και προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους Σύριους οι οποίοι φεύγουν από τη χώρα τους. Ε, πήγαμε στη Χατιλά την προηγούμενη εβδομάδα και είδαμε δύο καταβλισμούς εκεί προσφύγων και μου έκανε εντύπωση τι συνθήκες επικρατούν στον καταβλισμό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ακόμα και όταν οι συνθήκε είναι καλές, κάποιοι άνθρωποι μένουν εκεί δύο χρόνια πολλές φορές. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η διεθνή κοινότητα γενικότερα να στηρίξουν την Τουρκία στις προσπάθειες που κάνει για να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική διάσταση της Συριακής κρίσης. Είναι ζωτική σημασία λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία να καταλήξουν σε αμοιβαία κατανόηση προκειμένου να προσφέρουν την ανθρωπιστική βοήθεια που χρειάζεται. Πρόεδρε, η έκθεση καταδικάζει έντονα την ε, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας από το ΠΚΚ και θέλει να ενισχυθεί η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Προκειμένου να διευκολυνθεί μια τέτοια συνεργασία, η Τουρκία πρέπει να εγκρίνει ένα νόμο προστασίας δεδομένων και νομοθεσία επίσης για την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ώστε να καταλήξουμε και σε συμφωνία με την Europol και η, να υπάρξει έτσι και δικαστική συνεργασία και να γίνει σχετική υπογραφή με την Eurojust. Το θέμα, ε, το κουρδικό δεν έχει λυθεί και στην έκθεση ζητάει η Επιτροπή από όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συνεργαστούν για να ενισχυθεί ο πολιτικός διάλογος και να υπάρξει και μια διαδικασία ε, υπέρ της συμμετοχής των πολιτών κουρδικής προέλευσης στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας. Από συζητήσει με την τουρκική κυβέρνηση και τον Αμπτουλά ε, Οτσαλάν ε, συζητήσεις γίνονται αυτή την εποχή. Και χαίρομαι επίσης και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό για άλλη μια φορά για το γεγονός ότι το CHP, δηλαδή το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζει τις συνομιλίες αυτές. Και υπάρχει τώρα μια μοναδική ευκαιρία, ένα ανοιχτό παράθυρο για να γίνουν σημαντικά βήματα προκειμένου να λυθεί αυτό. Γίνεται επίση δουλειά και πάνω στο Σύνταγμα. Είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία και αυτή Η σχετική επιτροπή του τουρκικού κοινοβουλίου πρέπει να θεωρηθεί προκειμένου να συνεχίσει το έργο της προς την κατεύθυνση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα όπως είναι η διάκριση των εξουσιών, η σχέση ανάμεσα στο κράτος, την κοινωνία και τη θρησκεία, θεμελιώδη δικαιώματα για όλους τους πολίτες, όπως επίσης και η ιδέα της συμμετοχής όλων των πολιτών στην ε, ζωή της χώρας. Λυπούμε για την ε, στάση της Τουρκίας να απόσχει τους τελευταίους έξι μήνες κατά διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας από τις ε, εργασίες. Τώρα υπάρχει μια ευκαιρία. Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας την έχασε όμως την ευκαιρία αυτή η Τουρκία για να λυθεί το πρόβλημα εκεί. Αρνήθηκε η Τουρκία και αρνείται να εφαρμόσει ε, πλήρως τα όσα αναφέρει το ε, επιπρόσθετο πρωτόκολλο, κάτι το οποίο εμποδίζει τη συνέχεια των, ε, τη συνέχεια των ε, διαπραγματεύσεων και των συνομιλιών. Αυτά είναι τα κύρια θέματα που ήθελα να σας υπογραμμίσω. Θα βρείτε βέβαια όλες τις εξελίξεις στο γραπτό κείμενο, στην έκθεση και ζητάω από τους ε, φλεμόδους ε, συναδέλφους να κοιτάξουν λίγο την ε, μετάφραση στα Ολλανδικά. Σίγουρα τα Ολλανδικά δεν είναι τόσο καλά όσο θα έπρεπε να είναι, οπότε ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, λέω μιλήτρια. Ευχαριστώ κύριο Ρουμπιόλς παρακαλώ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Πρόεδρε, δεν το λέω έτσι για τους τύπους. Ειλικρινά ε, συγχαίρω την εισηγήτρια για την ε, έκθεσή της. Με κάθε ειλικρίνεια. Διότι διάβασα το σχέδιο έκθεσης προσεκτικά και πιστεύω ότι αποτελεί ένα πάρα πολύ καλό σημείο κίνησης για τις συζητήσεις μας. Έχω την αίσθηση ότι όσο περνάνε τα χρόνια η συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων εδώ ενισχύεται όσον αφορά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων. Δυστυχώς και για λόγους γνωστούς βέβαια, που δεν θα επαναλάβω, η διαδικασία προχωρά ιδιαίτερα αργά. Και το θέμα δεν είναι μόνο η επιτάχυνση της διαδικασίας. Το πρόβλημα είναι ότι η διαδικασία πρέπει να είναι θετική, δηλαδή τα πολιτικά αποτελέσματα να είναι θετικά όσον αφορά τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην είναι αντιπαραγωγικά. Να βοηθήσει η διαδικασία σε όλο και βελτιωμένη κατανόηση μεταξύ μας και σε μεταρρυθμίσεις όπως αυτές που γίνονται τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία και πάνε προς τη θετική κατεύθυνση. Ελπίζω το 2013 να είναι ένα πιο θετικό έτος υπό αυτή την έννοια. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι θα γίνει αυτό. Το πρώτο είναι η κατάσταση στην ε, περιοχή. Αναμφίβολα πρέπει να υπάρξει όσο γίνεται μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ε, στην περιοχή, το ανθρωπιστικό. Δεύτερον, έχουν γίνει αλλαγές σε διάφορες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Γαλλία για παράδειγμα. Ο πρόεδρος Ολάντ ε, αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα και έχω την αίσθηση ότι υπάρχει κάποια αλλαγή. Δηλαδή οι αντιρρήσεις, οι πιο ουσιαστικές, οι πιο θεμελιώδεις που υπήρχαν από τον προηγούμενο πρόεδρο έχουν δώσει τη θέση τους σε μια πιο πραγματιστική στάση αξιολόγησης των πολιτικών και οικονομικών κριτηρίων για την ένταξη της Τουρκίας. Τώρα έχουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Επιτρόπου Φούλε, που θέλει να προχωρήσουμε βάσει μιας θετικής ημερήσιας, ε, ε, ε διάταξης που δεν αντικαθιστά βέβαια τις διαπραγματεύσεις, αλλά αποτελεί ένα στοιχείο δυναμισμού της διαδικασίας και ενισχύει τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Οι τουρκικές αρχές, κάποιες τουλάχιστον, είπαν ότι το 2023, 100 χρόνια δηλαδή από τότε που υπάρχει η τουρκική δημοκρατία, η Τουρκία πρέπει να είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν είμαι σε θέση να κάνω προβλέψεις χρονολογικού τύπου, αλλά βλέπω ότι ο στόχος να συνεχίσουμε, να βελτιώνουμε, να επιταχύνουμε, να κάνουμε πιο συγκεκριμένες τις διαπραγματεύσεις εν ώψη της ένταξης της Τουρκίας είναι μια δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και χρόνια. Υπάρχουν διάφορα ε, σημεία πάνω στο οποία θα επιμείνει η ομάδα μας. Βάσει πάντα μια θετική αξιολόγηση, έτσι που κάνουμε στην έκθεση. Κάποια τα ανέφερε η συνάδελφος από το ΕΛΚ πριν από λίγο. Το άνοιγμα νέων κεφαλαίων των σχετικών ιδιαίτερα με τη δικαιοσύνη, τα κεφάλαια δηλαδή 23 και 24. Έτσι όπως έχει κατάσταση σήμερα στην περιοχή, το κεφάλαιο 30 που αναφέρεται στις εξωτερικές σχέσεις θα μπορούσε να ήταν μια δυνατότητα επίσης πρέπει να στηρίξουμε και τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων. Πάντα όμως στη βάση του ότι υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες για μας είναι απαράδεκτες. Όπως για παράδειγμα το θέμα της ε, μη πλήρους ελευθερίας του λόγου. Έπειτα, το θέμα των νόμων των αντιτρομοκρατικών και το πόσο ευρύς είναι. Από την άλλη μεριά πιστεύουμε ότι είναι θετικό το ότι αρχίζουν οι συνομιλίες για να προχωρήσουμε σε λύση του κουρδικού, που σημαίνει αναγνώριση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των Κούρδων. Τέλος, ο πλουραλισμός μάλλον όσον αφορά την ε, συνένεση για ένα νέο σύνταγμα είναι επίσης ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση αυτή. Και είναι πολύ σημαντικό ε, για όλες τις ομάδες πιστεύω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλος, το Κυπριακό. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φροντίσουμε να μην ε, μπλέξουν τα πράγματα ακόμα περισσότερο, να βοηθήσουμε τις διαδικασίες διαπραγματεύσεων για να προχωρήσει αυτό το θέμα. Είναι ένα εμπόδιο το οποίο πιστεύουμε ότι μπορεί κάποια στιγμή να πάψει να υπάρχει για να βρει το δρόμο της προς την Ευρώπη η Τουρκία. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Νέης, έχει τώρα το λόγο. Uh, Mr. President. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι εδώ ο σκιώδης μας, ο Αλεξάνδρ Γκραφ Λάμσδορφ, γι' αυτό ε, θα κάνω εγώ κάποιες πρώτες παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο έκθεσης. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τη συντάκτρια, την εισηγήτρια, γιατί είναι εξαιρετικό το κείμενο, είναι ολοκληρωμένο, πλήρες, με αποχρώσεις, αντικειμενικό και αποτελεί νομίζω εξαιρετική βάση για να συνεχίσουμε να ε, το βελτιώνουμε και να βελτιώνουμε θεωρώ και τις σχέσεις μας με την Τουρκία και τους, Τουρκικού, τους Τούρκους βουλευτές ε, και τους ε, ε για τη διαμόρφωση της κοινή γνώμης. Τώρα, κάποια θετικά σημεία που θέλω να αναδείξω. Εκτιμώ ιδιαίτερα τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το Κυπριακό στην παράγραφο 23 με τρόπο ισορροπημένο, καταδείχνει ένα πιθανό δρόμο πρόοδου και αυτό είναι σημαντικό. Επίσης, είναι σημαντικό πιστεύω ότι δύο παραγράφους παρακάτω, στην παράγραφο 25, αναφέρεται η ουσία του προβλήματος σε σχέση με τις τριμερείς σχέσεις Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Τουρκία και άλλους. Εκεί διατυπώνεται η ουσία της σχέσης αυτής της τριμερούς με πολύ σαφή τρόπο. Νομίζω πέρσι ή πρόπερσι ε, που προσπαθήσαμε να κάνουμε ακριβώς αυτό και η Επιτροπή απέρριψε την τροπολογία μας ε, στο ψήφισμα τότε. Τώρα νομίζω ότι σαφέστατα εντοπίζουμε τα προβλήματα και άρα και την πιθανή λύση τους. Και προφανώς όσο ομάδα ελπίζουμε ότι θα είναι δυνατόν να συνεχιστεί να συνεχίσουμε τον πολιτικό διάλογο μεταξύ της τουρκικής κυβέρνησης από τη μία πλευρά, να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ ε, τουρκικής κυβέρνησης και των ε, ηγετών των Κούρδων, γιατί μετά από τόσες αιματοχυσίες και θύματα είναι πλέον ξεκάθαρο ότι κάτι θετικό μπορεί μόνο με πολιτικά μέσα και όχι με τη βία να επιτευχθεί. Φοβούμε ότι οι τρεις τελευταίες δολοφονίες των, των τριών γυναικών των ακτιβιστριών του ΠΚΚ στο Παρίσι είναι μια προσπάθεια, μια απόπειρα εκτροχιασμού των συνομιλιών. Άρα, τόσο πολύ περισσότερο πρέπει να χαιρετήσουμε το γεγονός ότι είναι αποφασισμένη η Τουρκία να συνεχίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μέχρι σότου, όπως ελπίζομαι, καταλήξουν σε θετικό αποτέλεσμα. Τέλος, στηρίζομαι την έκκληση στην έκθεση αυτή προς τα 27 κράτη-μέλη να ανοίξουν τα κεφάλαια 23 και 24. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε ότι ενώ εγκρίθηκε να, να γίνει αυτό προς το Μαυροβούνιο ε, υπάρχει άρνηση να γίνει προς την Τουρκία γιατί είναι μια ε, χώρα σεβαστή το Μαυροβούνιο βεβαίως ε, είναι σημαντική για μας και μετά το διαμελισμό της ε, Ιουγκοσλαβίας, μετά τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας ε, όλες ε, οι χώρες που δημιουργήθηκαν, οι καινούριε χώρες ε, δικαιούνται ένα ειρηνικό μέλλον. Η Τουρκία όμως είναι μια μείζον χώρα, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά παγκοσμίω. Και αν δούμε τι συμβαίνει δυστυχώς στην Συρία και στην άμεση γειτονία της, βλέπουμε ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό η σχέση με την Τουρκία να αναπτυχθεί με τρόπο θετικό σε υγιή βάση. Και γι' αυτό στηρίζουμε την έκκληση στα κράτη-μέλη να αφήσουν να ανοίξουν τα κεφάλαια 23 και 24, πόσο μάλλον που τόσο πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιμένουν για τις ε, αναγκαίες βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν σε όλους αυτούς τους τομείς που καλύπτουν τα κεφάλαια αυτά. Γιατί να μην ανοίξουν λοιπόν. Και πάλι ε, σας είπα δεν είμαι σκιώδης εισηγήτρια και δεν ξέρω αν θα υποκαταθέσουμε τροπολογίες, αλλά συνολικά και εγώ και η, και η ομάδα μου θεωρούμε την έκθεση εξαιρετική και προσβλέπουμε σε περαιτέρω εξελίξεις. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Αλαβράκος παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ειλικρινώς θέλω να συγχαρώ την κυρία Όιμιν Ρόιτιν διότι για τρίτη ή τέταρτη χρονιά μας παρουσιάζει μια σοβαρή και ισορροπημένη έκθεση και μπορώ να πω ότι η κυρία Ρόιτεν με έχει πείσει ότι είναι ειδική περί τα τουρκικά θέματα περισσότερων παντός άλλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσωπικά πιστεύω ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, έχει διεθνές κύρος και Επιτρέψτε μου να πω ότι θεωρώ την παρούσα πολιτική της ηγεσία μία από τις καλύτερες πολιτικές ηγεσίες τις οποίες είχε στα τελευταία χρόνια. Παρακολουθώ ιδιαίτερα τη συμπεριφορά της στις τρέχουσες εξελίξεις στη Συρία και με ικανοποιεί ιδιαίτερο η δειλή έστω διαπραγμάτισή της και το άνοιγμα που κάνει στο κουρδικό θέμα. Θεωρώ όμως ότι η Τουρκία δεν συμπεριφέρεται με την σύνεση που της αναλογεί σαν κράτος κύρους σε σχέση με το Κυπριακό. Έτσι συμφωνώ απόλυτα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 22 της εκθέσεως για τη διακοπή των διπλωματικών επαφών της Τουρκίας με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, αφού η κίνηση αυτής της Τουρκίας, καθώς και πολυάριθμες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων σχετικά με αυτό, δεν βοηθά στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών, ενώ αποτελεί ενδεικτικό της άρνησης της Τουρκίας να συνεργαστεί με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σεβαστεί τις ευρωπαϊκές αξίες. Οι σχέσεις με τα γειτονικά κράτη δεν μπορώ να πω ότι βρίσκονται στο καλύτερο σημείο το οποίο θα είναι το επιθυμητό διότι παρά τις συνεχές προτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σχέσεις καλής γειτονίας και ειρηνικής διευθέτησης των προβλημάτων, η Τουρκία εξακολουθεί να προβαίνει σε απειλές εναντίον γειτονικών κρατών και να προβάλλει βέτο στη συμμετοχή ευρωπαϊκών κρατών μελών σε διεθνείς οργανισμούς όπου συμμετέχει. Χαρακτηριστικά η Τουρκία παρεμπόδισε την περασμένη Τρίτη την είσοδο της Κύπρου και του Ισραήλ στο Συμβούλιο της Διεθνούς Υπηρεσίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το ΙΡΕΝΑ. Η Τουρκία ήταν η μόνη μεταξύ των 185 χωρών μελών που αντιτάχθηκε στις δύο υποψηφιότητες. Πέρα από το κάζους μπέλη κατά της Ελλάδος, έχει ήδη αυτό από το 1995 αποτελέσει απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, το οποίο αρνείται να το αποσύρει. Επιπλέον τούτου, η Τουρκία απειλεί με θερμό επεισόδιο σε περίπτωση που η Ελλάδα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά τη που απορρέει από τι διεθνεί συμβάσει του ΟΗΕ, ω προ το δικαίωμα κάθε κράτου για ανακήρυξη αποκλειστική οικονομική ζώνη. Μερικοί διαπίστωσα ότι αυτή τη χρονιά δεν περιλαμβάνεται στην έκθεση καμία αναφορά στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο τη θάλασσα που εξακολουθεί να αρνείται να υπογράψει η Τουρκία. Θέλω να πιστεύω ότι ε, η έκθεση της κυρίας ε, Ρόιτερ αποτελεί συνέχεια των εκθέσεων της εξυπαρχής και συνέχεια των λοιπόν ψηφισμάτων και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως πολιτικές διαπιστώσεις παρελθόντων ετών επί των οποίων δεν υπάρχουν εξελίξεις θεωρώ ότι εξακολουθούν εις το ακέραιο να ισχύουν και επομένως να χρήζουν απαντήσεις εκ μέρους της Τουρκίας. Παρά τις εγχώριες και διεθνείς επικρίσεις κατά της φυλάκησης και δίωξης των δημοσιογράφων στην Τουρκία, η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει αποφασιστικά. Είναι απαραίτητο η Τουρκία να σεβαστεί τις δημοκρατικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα αν θέλει να έχει μια ευρωπαϊκή πορεία. Σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων, η ελευθερία του τύπου στην Τουρκία συστηματικά καταστέλλεται ενώ η τελευταία κατέχει την υψηλότερη θέση παγκοσμίω ως προς τον απόλυτο αριθμό των κρατουμένων δημοσιογράφων. Οι τουρκικές αρχές πρέπει να δείξουν πνεύμα συνεργασίες και η Τουρκία να συμμορφωθεί ως προς τις υποχρεώσεις της έναν των μεταναστών και των ετούντων άσυλο. Χαιρετίζω την πρόταση της συγκητρίας που παροτρύνει την Τουρκία να υπογράψει και να εφαρμόσει τη Συμφωνία Επανεισδοχής χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Και στο σημείο αυτό θέλω να πω τα εξή θέλω να πω ότι πέραν από τον εξευρωπαϊσμό υπάρχει η παγκοσμιοποίηση, την οποία πολλά κράτη, ιδιαίτερα τις περιοχές των Βαλκανίων, δεν την έχουν αντιληφθεί. Ο κόσμος γίνεται ένας. Μοιραία σε κάποια στιγμή θα υπάρχει συναδέλφωση εντός εισαγωγικών ή συνεργασία των λαών σε επέκεινα στάδιο αυτού που υπάρχει. Επομένως εκείνο το οποίο προέχει στις παρούσες φάσεις και εν ώψη των εξελίξεων που τις βλέπουμε ορατές θα είναι πιο Να διατηρήσουμε τις καλές σχέσεις ο ένας με τον άλλον και να μην ανταλλάσσει ο ένας με τον άλλον απειλές ή εκφράσεις που δεν θα διευκολύνουν τη ζωή του στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Και η κυρία Λούνατσεκ τώρα ε, για τους, την ομάδα των Πρασίνων και σε τον γύρο των σκιωδών εισηγητών. Η κυρία Λούνατσεκ, παρακαλώ. Καλώς. Δεν με πειράζει να μιλήσει πρώτος ο κύριος ε, Τάνοκ, γιατί εγώ εκπροσωπώ την κυρία Φλότρ που δεν μπόρεσε να έρθει λόγω του χιονιού, ε, οπότε Εξ του Τζέφρι Βαν Όρντεν που είναι σκιώδης θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Όμεν Ρόιτεν για εξαιρετική και συνεκτική έκθεση. Ειλικρινώς πολλά επαναλαμβάνονται από τα προηγούμενα χρόνια. Είναι παρόμοια η κατάσταση εδώ και δύο-τρία χρόνια στην εξωτερική πολιτική, μιλάμε όμως για το ΜΙΝΤ, είχαμε παλιά το BRICS, δηλαδή Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, τώρα έχουμε το Μεξικό, Ινδονησία, Νιγηρία και Τουρκία, το ΜΙΝΤ, που είναι οι αναδυόμενες μεγάλες οικονομίες της επόμενης τρίκοντα αιτίας. Οπότε η Τουρκία είναι αναδυόμενη και στρατιωτική αλλά και οικονομική δύναμη. Και ό,τι και να πιστεύει κανείς για την ένταξη της Τουρκίας, ε, προφανώς ε, είναι ένας πολύ ισχυρός, ε, σημαντικός παγκόσμιος παίκτη και η υποψηφιότητά της στην Ευρώπη βραδιπορεί λόγω των πολλών προβλημάτων που αναφέρονται εδώ και αναφέρθηκαν και παλιότερα και προέρχονται από τη μη εφαρμογή του πρωτοκόλου της Άγκυρας και ιδιαίτερα τη μη αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, το θέμα της του το βέτο στη συνεργασία ε, με τον ΝΑΤΟ ε, και την ένταξη της Κύπρου την ε, Ανατολική Μεσόγειο όπου η Τουρκία δραστηριοποιείται και η Κύπρος δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τους πόρους της λόγω της μη αναγνώρισης της ΑΟΖ. Επίσης το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φυλάκιση δημοσιογράφων, ιδιαίτερα από την κουρδική μειονότητα και Κούρδους ε, ε, πολιτικούς από την τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης υπάρχουν και θέματα ε, θρησκευτικών μειονοτήτων. υπάρχουν ε, μειονότητες επίσης το θέμα του, της σχολής της Χάλκης Επίσης, ε, κάτι καλό είναι ο διάλογος που ανακοινώθηκε μεταξύ της τουρκικής κυβέρνησης και του Αμπτουλάου Τσαλάν. Δεν ε, ε, ξέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις τρομοκρατικές δραστηριότητες των Κούρδων μετά από την φυλάκιση του Τσαλάν. Πάντως αναγνωρίζεται τώρα το κουρδικό, αναγνωρίζεται ότι πρέπει να βρεθεί πολιτική λύση και βέβαια ε, ήταν ε, πολύ δυσάρεστο το ήταν πάρα πολύ ε, τραγική η δολοφονία αυτή. ελπίσουμε ότι δεν θα εμποδίσει τις περαιτέρω ε, συνομιλίες, τις ειρηνευτικές. Επίσης ε, θα πρέπει να υπάρξει στη Συρία ε, μια μετάβαση ομαλή στην ε, δημοκρατία. Εδώ έπαιξε ρόλο θετικό η Τουρκία, ε, όπως και απέτρεψε το να πλησιάσει τη Συρία το Ιράν. Επίσης χαιρετίζω το... Επίσης καταδικάζω το γεγονός ότι παραμένουν κλειστά τα σύνορα με την Αρμενία. Είναι... θα ήταν πολύ σημαντικό να αναγνωρίσει η Τουρκία ότι δεν οδηγεί πουθενά αυτό. Ε, το μόνο που επιτυγχάνει είναι να διατηρεί την πόλωση στα ανατολικά σύνορα. Ε, καλό θα ήταν φέτος να υπάρξουν κάποια εισιδήσεις προς θετική κατεύθυνση. Ε, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την προσχώρηση της Τουρκίας, αλλά προφανώς θα πρέπει να ε, παίξουμε επικοδομητικό ρόλο αφού είναι μεγάλη δύναμη η Τουρκία, ε, είναι σημαντικός οικονομικός και εμπορικός εταίρος και είναι σημαντικό να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας ε, και βελτιώνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το μποϊκοτάζ της Τουρκίας στην Κυπριακή Προεδρία βέβαια δεν βοήθησε καθόλου και αυτό είναι λυπηρό. Όμως υπάρχουν και κάποια θετικά Αναφέρθηκα ήδη στις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Κουρδικό. Συνολικά Πάλι θέλω να συγχαρώ την συγγήτρια, είναι πολύ περιεκτική έκθεση επί ενός ε, θέματος περίπλοκου και με πολλές λεπτομέρειες ε, ένα πολιτικό θέμα που απασχόλησε τα τελευταία χρόνια την ομάδα μου ε, γιατί το θεωρούμε προτεραιότητα. Επίσης, τα κεφάλαια 23 και 24 συστήνουμε να μελετηθούν, γιατί θέματα εσωτερικών υποθέσεων, καταπολέμηση διαφθοράς, ε, οργανωμένου εγκλήματος. Παραμένουν πολύ σημαντικά θέματα προκειμένου να πείσουμε και του εκλογείς μα εμεί στην Ευρώπη ε, υπέρ της ένταξης της ε, Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα θα πρέπει να δούμε το θέμα της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, γιατί αυτό απασχολεί και θα απασχολεί πολύ τους πολίτες μας κατά την προσχώρηση της χώρας αυτής. κυρία ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Τώρα θα ήθελα να μιλήσω για την κυρία Φλότρ, τη σκιώδη ηγήτριά μα, η οποία παγιδεύτηκε από τα χιόνια όπω και πολλοί άλλοι και δεν ήρθε έγκαιρα. Εξ ονόματος της Ελένη Φλότρ και της ομάδας μου, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Όμεν Ρόιτεν για την πολύ ισορροπημένη και καλή έκθεση ε, που στηριχθήκε σε καλή συνεργασία των ε, σκιωδών εισηγητών. Ε, υπάρχουν θετικά σημεία που θέλω να αναφέρω στην έκθεση. Όπως είπε η κυρία Όμεν εδώ υπάρχει το αίτημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνολικά να ανοίξουν τα κεφάλαια 23 και 24. Επίσης, το γεγονός ότι η κυρία Ομεν στην έκθεσή της έχει συμπεριλάβει το ότι ε, τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ θα πρέπει να διασφαλίζονται και το αίτημα έκκληση περισσότερο προς την Τουρκία και την Κύπρο να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες προς την κατεύθυνση συμβιβαστικής λύσης. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για να προχωρήσουμε. Επίσης θέλω να αναγνωρίσω το ρόλο που παίζει η Τουρκία στην ανθρωπιστική κρίση της Συρίας και γύρω από τη Συρία και πώς αντιμετωπίζει τον ε, μεγάλο αριθμό προσφύγων που υποδέχθηκε. Είναι καλό που υπάρχει στην έκθεση. Υπάρχουν ορισμένα θέματα που θα θέλαμε να βελτιώσουμε από τη δική μας την πλευρά και γι' αυτό θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες. Αναφέρομαι σε ορισμένα θέματα. Πρώτον, είναι καλό ότι υπάρχουν κάποιες αναφορές στο οικολογικό και ενεργειακό δυναμικό της χώρας. Αλλά είναι μικρή αναφορά στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Εδώ θα θέλαμε μια ευρύτερη ανάλυση των σημείων και θα θέλαμε να επισέλθουμε στο θέμα των πυρηνικών εργοστασίων που σχεδιάζονται εκεί και ποιο είναι το δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Τουρκία, γιατί δεν αξιοποιούνται πολύ. Προσθέτω εν παρόδο ότι βρίσκουμε πολύ θετικό το γεγονός ότι το Διοικητικό Δικαστήριο της Τουρκίας πρόσφατα ε, σταμάτησε την κατασκευή ε, του φράγματος που δεν πληρούσε περιβαλλοντικά κριτήρια. Ε, ξαναγυρίζω στο θέμα των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Εμείς θα θέλαμε να ζητήσουμε το κεφάλαιο απασχόληση και κοινωνικά θέματα να ανοίξει με την χώρα αυτή, γιατί τα δικαιώματα των συνδικαλιστών στην Τουρκία δεν γίνονται σεβαστά όπως πρέπει και αυτό θα θέλαμε να συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας όπως και η τήρηση των προτύπων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Και αυτό είναι πολύ κεντρικό θέμα. Ε, ένα άλλο θέμα που έθιξαν και άλλοι συνάδελφοι είναι η σχέση των ε, Κούρδων ε, και την, της ειρηνευτικής διαδικασίας, η ειρηνευτική διαδικασία που τώρα γίνεται μεταξύ τουρκικής κυβέρνησης και ΠΚΚ Τσαλάν. Νομίζω ότι είναι θετικό να χαιρετήσουμε αυτή τη διαδικασία ως Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως βρίσκω ότι είναι απαραίτητο και θα κατατεθεί σχετική τροπολογία από εμά να επικρίνουμε τους νόμους κατά της τρομοκρατίας που περιορίζουν πολύ την ελευθερία έκφρασης θα, θα καταθέσουμε σχετική τροπολογία. Επίσης θέλω να καταγραφεί και στην Επιτροπή μας ότι ελπίζομαι ότι η ε, η άγρια εκτέλεση των τριών ακτιβιστριών στο Παρίσι δεν θα εμποδίσει τις ειρηνευτικές διαδικασίες τουρκικής κυβέρνησης και Κούρδων. Τουλάχιστον ε, αυτό το θέμα πρέπει να το και, θα πρέπει να πάνε στα δικαστήρια ε, της γαλλικής δικαιοσύνης οι ένοχοι. Επίσης ε, ε, η Πίνα Σέλικ είναι μια ε, κοινωνιολόγος ακτιβίστρια η οποία ήταν στο Στρασβούργο, δικάζεται και την είδαμε, τη συναντήσαμε ορισμένοι από εμάς. Ελπίζω στις 24 Ιανουαρίου που θα εκδικαστεί η υπόφαση να αθωωθεί. Και, και βέβαια αν ο Μιγέννη το καταδικαστεί θα πρέπει αυτό να αναφερθεί στην έκθεση. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Όμουν Ρόιτερ. Σας ευχαριστώ πολύ. 11 ομιλητές έχουμε τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσπαθήσετε να περιορίσετε τις παρεμβάσεις σας στα δύο λεπτά. Ο πρώτος που θα το προσπαθήσει είναι ο κύριος Γκρέαμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να καλωσορίσω την έκθεση, αλλά για να μην σπαταλώ το χρόνο της Επιτροπής θα μείνω σε κάποια περιορισμένα θέματα, γιατί η κυρία Νέιτ έδωσε το στίγμα της ε, ομάδας μας. Θα ε, ήθελα να μιλήσω για εκείνα τα κομμάτια της έκθεσης που μιλάνε για την ενέργεια. Η κυρία Όμεν Ρόιτεν εντοπίζει ο δυναμικό της ε, Τουρκίας να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων και των οδών μεταφοράς της ενέργειας καλωσορίζει τη συνεργασία ε, της Τουρκίας για τα ενεργειακά θέματα. Είναι όντως ένα ζήτημα ε, Όλα ένα και μεγαλύτερη σημασία δεδομένη της επικίνδυνης εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η ομάδα μου καλωσορίζει την αυξημένη συνεργασία, τη συμφωνία μάλλον ε, αυξημένης για την ενέργεια του Στουτγκάρδη στο περασμένο Ιούνιο. Θα θέλαμε να γίνονται περισσότερα όσον αφορά τις υποδομές και την ευφυή ανάπτυξη και πιστεύουμε πως η συνεργασία Ένωσης με την Τουρκία στα θέματα της ενέργειας θα πρέπει να είναι περισσότερο από ότι απλά η ενέργεια. Θα πρέπει να μοιράζονται οι πόροι, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ανανεώσιμες για τις οποίες μίλησε και η κυρία Λούνατσεκ. Ε, θα τίνουμε να βλέπουμε την Τουρκία ως ένα κόμβο, αλλά κυρίως σε σχέση με το φυσικό αέριο. Αυτό πρέπει να αλλάξει και η ομάδα, η παρακολούθηση πρέπει να συναντιέται πιο πολύ από ό,τι μια φορά το χρόνο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να αποτελέσουν κλειδί της σχέσης ανάμεσα στην Ένωση και την Τουρκία και να συμπεριληφθεί και η ανάπτυξη νέων πράσινων αποτελεσματικών ενεργειών στην Τουρκία, που η Τουρκία τώρα προετοιμάζει γύρω στα 50 ε, στις 50 εγκατοστάσεις ε, που θα λειτουργούν με άνθρακα. Εμείς θα πρέπει να προσβλέπουμε στη σύνδεση της Τουρκίας με ένα μεγαλύτερο μείγμα, πλέγμα ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και προς τα εκεί θα πρέπει να την παροτρύνουμε. Εάν δεν ενδιαφέρονται οι συνάδελφοι, εγώ διοργανώνω σεμινάριο αύριο από τις 4 μέχρι τις 6.30 στην αίθουσα 1G2 που είναι ακριβώς κάτω από το την εδώ για την ε, συνεργασία για την ενέργεια με την Τουρκία. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Κοπά, δύο λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τη Ρία Ομενρόιτεν για αυτό το σχέδιο που μας δίνει μια σπουδαία βάση για συζήτηση στην Επιτροπή αυτή. Κατανοώ απόλυτα τις δυσκολίες της εισηγήτριας των να όλα αυτά τα θέματα που προκύπτουν από τις σχέσεις μας με την υποψήφια χώρα. Ε, σε ένα μόνο σχέδιο. Γνωρίζει βεβαίως ότι αυτό σημαίνει περισσότερες τροπολογίες από ό,τι συνήθω και εγώ είμαι πρόθυμη να περιοριστώ στα απολύτως απαραίτητα και προσβλέπω στην συνεργασία μας. Όπως είναι γνωστό δυστυχώ, οι σχέσει ενωσής με την Τουρκία ε, ε, περνάνε μια περίοδο τελμάτωση περιμένουμε ένα μήνυμα και από την πρώτη παράγραφο ε, εσείς συγχαίρετε την ε, Τουρκία για την εφαρμογή της θετική ε, ατζέντα και συντονίζει την στρατηγική της σημασία. Αυτό όμω δεν πρέπει να σκιάζει την πραγματικότητα και την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων. Θα ήθελα, σε... δεν θέλω εδώ τώρα να μιλήσω για ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα, όπου η κατάσταση διαρκώ επιδεινώνεται, ότι πολλοί συνάδελφοι ήδη το ανέφεραν. Κατά τη, μου, κατά τη γνώμη μου, οι τελευταίοι μήνες έχουν δείξει σαφώς ότι η Τουρκία συνεχίζει, αντιλαμβάνεται μάλλον τις σχέσεις της με την Ένωση, ε, γιατί μόνο όταν προωθούνται οι προτεραιότητες της Άγκυρας και η χώρα έχει παγώσει τις σχέσεις της με την κυλιόμενη Προεδρία της Ένωσης. Η Τουρκία εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να αγνοεί και να παρακάμπτει την Κυπριακή Προεδρία χωρίς συνέπειες. Γι' αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε στην έκθεση ότι τέτοια ε, λαφριά προσέγγιση και αλακάρτ ε, δεν είναι αποδεκτή από το Ευρωκοινοβούλιο. Να θυμίσω δε στην Επιτροπή ότι η επιμονή των Τούρκων ομολόγων μας που είναι πρόσδεκτοι εδώ, ε, που είναι βουλευτές από την Εθνοσυνέλευση, δεν δέχονται την παρουσία ενός εκπροσώπου της Κυπρικής Προεδρίας και αυτό οδήγησε σε ακύρωση της 17ης ε, συνεδρίασης της Μικτής ε, Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής. Α, είναι παράγραφο 22. Ήδη αναφέρατε. Ναι, ναι, το ξέρω. Το είδα. Διακόψη κυρία Μενρόιτεν. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί αυτό στο τομέα της έκθεσης που, λέγεται, που τιτλοφορείται «Επικοδομητικός διάλογος και κοινή συνεννόηση». Όντως υπάρχει αναφορά σε αυτή την τουρκική στάση στην παράγραφο 22 υπό τον τίτλο «Καλές σχέσεις για την ίαση». Η εντύπωσή μου είναι πως δεν είναι ακριβέστερη αυτή η επιλογή γιατί δεν είναι θέμα ε, καλής γειτονιασής ανάμεσα στην Τουρκία και την Κύπρο είναι θέμα αρχής και σεβασμού για τις ευρωπαϊκές συνθήκες και την θεσμική τάξη από μια υποψήφια χώρα. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα τμήμα που αφιερώνεται στην ανάγκη δημιουργίας οικοδομητικού διαλόγου χωρίς να αναφερόμαστε σε αυτά τα προβλήματα. Μιλώντα τώρα για τι καλέ σχέσει γετνίαση, επιπλέον τα προβλήματα δεν περιορίζονται στο Κυπριακό. Το 2012 είχαμε διαπιστώσαμε τη συνέχιση των σκλημάκωσης των τουρκικών απειλών που ανοιχτά προκαλούν τα κυρίαρχα δικαιώματα ε, κρατών μελών και παραβλέπουν τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου. Δύο τίτλοι ακόμα και θα έχω τη δυνατότητα μέσω των τροπολογιών μου να επεκταθώ. Καταρχήν, συμφωνώ με τους συναδέλφους για το θέμα της δολοφονίας των τριών Κούρδων γυναικών στο Παρίσι και επίσης συμφωνώ με την κυρία Λούνατζη για το θέμα της Πινάρ Σαλέκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Σκούτ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα και εγώ ευχαριστώ πολύ τη Ρία, την εισηγήτρια, για την εξαίρετη και ισορροπημένη της έκθεση. Είναι πράγματι πολύ καλό να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που θα θέλαμε είναι όθεση της διαδικασίας και το λέει αυτό η έκθεση. Είμαστε σε μια πολύ σημαντική διαδικασία, το βλέπουμε αυτό στην Τουρκία και για το κουρδικό και υπάρχουν ένα σωρό θέματα που μένουν ακόμα να λυθούν όπως η ελευθερία της έκφρασης. Συμφωνώ με τη Ρία ότι το σημαντικό είναι να ανοίξουν τα κεφάλαια 23 και 24 όχι μόνο για την ελευθερία του τύπου, γενικότερα για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και όσον αφορά τη βία σε βάρος των γυναικών είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να λυθεί. Και μόνο έτσι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Το τέταρτο πακέτο για την ε, δικαιοσύνη και τις μεταρρυθμίσεις επίσης είναι πολύ σημαντικό. Η δουλειά που γίνεται για τη μεταρρυθμίση στο Σύνταγμα. Και το τελευταίο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πως και εδώ πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις όταν επιστρέφει ο κόσμος στην Τουρκία ότι τα θεμελιώδη του δικαιώματα θα προστατεύονται. Τέλος, τέλος, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε και η Ρία όσον αφορά την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με τους πρόσφυγες από την Συρία. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Σοφοκλέους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και οφείλω να παραδεχτώ ότι καταβάλλεται προσπάθεια να παρουσιάσει μια ισορροπημένη έκθεση. Όμως το μεγάλο ερώτημα προσωπικά εκτιμώ είναι όχι το τι επέτυχε μέχρι σήμερα η Τουρκία, αλλά τι όφιλε να πράξει μέχρι σήμερα και δεν το έπραξε. Κατά καιρού δυστυχώς επαναληπτικά προσβάλλει θα τολμήσω να πω εκβιάζει με δηλώσεις εξωματούχων της την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα επί της ουσίας, η Τουρκία συνεχίζει να καταπατεί και να παραβιάζει κατάφορα όλα τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, την διεθνή ένωμη τάξη και να μην σέβεται τις αρχές της ιδίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού έδαφος της συνεχίζει να βρίσκεται υποστρατοτική κατοχή. Αναφορικά με τα ενταξιακά κεφάλαια 15, 23, 24, αποτελεί πρόκληση να επιδιώκεται το άνοιγμά τους αφού δεν έχει προχωρήσει η ενταξιακή πορεία και η ίδια η Τουρκία δεν φαίνεται πρόθυμη να κάνει υποχωρήσεις για να συνεχιστούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Σωστά αναφέρεται στην έκθεση ότι η Κυπριακή Προεδρία δεν αξιοποιήθηκε από την Τουρκία όπως θα έπρεπε και χάθηκε μια σημαντική ευκαιρία την εξομάλυση των σχέσεων των δύο χωρών. Συγκεκριμένα, συνεχίζεται ο παράνομος επικισμός που στόχο έχει την δημογραφική αλλαγή του νησιού. Παραμένει αδιευκρίνηστη η τύχη των αγνωμένων λόγω της άρνησης Τουρκίας να συνεργαστεί με την Κυπριακή Δημοκρατία. Συνεχίζεται η στρατοτική κατοχή και ο διαμελισμός μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος η Τουρκία απειλεί την Κύπρο λόγω της έρευνας που γίνεται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του νησιού με στόχο την εξόριξη φυσικού αερίου. Ως εκ τούτου, συμπερασματικά, δεν συμφωνούμε με την εισήγηση για άνοιγμα των κεφαλαίων 15, 23 και 24. Ευχαριστώ. Thank you very much. Mr. Angourakis, Ο κύριος Αγκουράκης. Κύριε Πρόεδρε, ε, καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω και εγώ τους εκπροσώπους του τουρκικού λαού, μεγάλος λαός, μεγάλη χώρα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ξέρω ότι το κόμμα μου είναι αντίθετο με την ένταξη της ε, Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θεωρούμε ότι αυτό θα οξύνει πάρα πολύ τα προβλήματα των εργαζομένων εκεί. Πάντω ε, δεν θα χρησιμοποιήσω τον χρόνο μου για το ζήτημα αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει μια άλλη ευκαιρία. Θα ήθελα να επικεντρωθώ κυρίω στο θέμα του Κυπριακού και να κάνω μια παρατήρηση όσον αφορά το θέμα τη Συρία. Εντελώ αρνητική θεωρώ την ε, πολιτική τη τουρκική κυβέρνηση στο θέμα τη Συρία. Έχει μεγάλη ευθύνη για, τα, ε, για το δράμα του Συριακού λαού και πολύ περισσότερο θεωρώ εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη την τοποθέτηση των πυράβλων Patriot στο έδαφος της, Συρίας, ε, της ε, Τουρκίας, στα σύνορα με τη Συρία, μια κατάσταση η οποία θα επιδεινώσει την κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό και η αναφορά στην έκθεση που συζητάμε σήμερα είναι στο σημείο 23, ε, νομίζουμε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές παραλήψεις οι οποίες δεν πρέπει να τις δεχτούμε, αλλιώνουν εντελώς και το πνεύμα ε, παλιότερων ε, κειμένων του, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εξελίξεων. Πρώτο ζήτημα, εκεί που γίνεται λόγος για το θέμα της επανένωσης της Κύπρου, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι η επανένωση πρέπει να γίνει στη βάση των αποφάσεων του, του ΟΗΕ και των ε, αποφάσεων υψηλού επίπεδου του 1977 και του 1979 στη βάση μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην υπάρχουν παρερμηνίες, για να μην ε, ε, και για να προχωρήσει η διαδικασία. Δεύτερο ζήτημα, πάλι για το θέμα του Κυπριακού, εκεί που γίνεται λόγος για, την επανέναρξη των ε, συνομιλιών και της διαδικασίας συνεννόησης, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια αναφορά που να τονίζει το πραγματικό γεγονός ότι παρά τις προσπάθειες που έκανε ο πρόεδρος Χριστόφιας, τόσο η Τουρκία όσο και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων δυστυχώς δεν επιτρέψαν στο να συνεχιστεί η διαδικασία συνεννόησης ε, ε, στην Κύπρο και έχουμε μάλιστα και μία ε, υποχώρηση από προηγούμενες συμφωνίες και προηγούμενα βήματα προς τα μπρος. Τρίτο ζήτημα όσον αφορά την αναφορά στην, στο απευθείας εμπόριο θεωρούμε ότι εδώ είναι σε λάθος θέση πολύ περισσότερο δεν υπάρχει και νομική βάση όσον αφορά τον ΟΗΕ και εν πάση περιπτώσει έτσι πως γίνεται αναφορά στο συγκεκριμένο σημείο ε, θα ε, επιτευχθεί ακριβώς το αντίθετο από αυτό που επιδιώκει η έκθεση, δηλαδή το να, ε, να ξεκινήσουν ξανά οι συνομιλίες, διότι ενισχύει το ψευδοκράτος στην Βορεια Κύπρο. Τέταρτο ζήτημα είναι το ζήτημα που έχει να κάνει με το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και την τοποθέτηση της Τουρκίας σε αυτό το ανεφέρετο δικαιώμα. Time, please, Mr. Time, time. Τελειώνετε παρακαλώ, τελείωσε ο χρόνος σας. Ε, I'm finished, Mr. President. is, ε, ε, μιλάω για το θέμα της, της ΑΟΣ και αν τελευταίο ζήτημα είναι για τους αγνοούμενους. Είναι η μοναδική περίπτωση όπου οι δύο κοινότητες συνεργάζονται και πρέπει η Τουρκία να επιτρέψει την συνέχιση των έρευνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Mrs. Theoharus, please. Η κυρία Θεοχάρους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα να καλωσορίσω την, τους α, Τούρκους συναδέλφους της Τουρκικής Συνέλευσης που βρίσκονται εδώ και αμέσως μετά να συγχαρώ την φίλη Ρία για την πολύ καλή και συνενετική έκθεση που έχει καταθέσει. Η έκθεση αυτή μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη αν δεχτεί η κυρία Όμεν και αν όλοι συμφωνήσουμε σε κάποιες α, αλλαγές και τροποποίησεις. Βεβαίως, τονίζεται ο όγκος των συναλλαγών και η δύναμη και η στρατηγική σημασία της Τουρκίας ε, στον κόσμο, αλλά εγώ σκεφτόμαι ότι η Ευρώπη δεν στήριζεται μόνο σε όγκους συναλλαγών και στρατηγικές σημασίες, αλλά σε αρχές, δημοκρατικές αξίες, ε, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς νόμου. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντα. Πρέπει να βοηθήσουμε την Τουρκία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέλουμε πάρα πολύ. Και εμεί ω μικρό και αδύναμο κράτο θέλουμε ένα ισχυρό δημοκρατικό γείτονα αλλά πρέπει και η ίδια η Τουρκία να βοηθήσει τον εαυτό της και την ενταξιακή της πορεία. Δεν θα μιλήσω για όλα τα άλλα τα οποία έχουν αναφερθεί από τους συναδέλφους για να κερδίσω λίγο χρόνο, παρόλο που θα ήθελα να μιλήσω αρκετή ώρα. Πρέπει όμως κατά την εκτίμησή μας να γίνει αναφορά, ρητή αναφορά για τις ευθύνε της Άγκυρας στη στασιμότητα όσον αφορά το Κυπριακό. Το Κυπριακό δεν είναι δικοινοτική διαφορά ή διαφορά εδαφική διασυνοριακή. Είναι θέμα στρατιωτικής κατοχής και αυτή τη στιγμή κατέχεται τμήμα του ευρωπαϊκού εδάφους από στρατιωτικές δυνάμεις της Τουρκίας. Πρέπει να γίνει αναφορά στην υβριστική συμπεριφορά απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία, απέναντι στην Κυπριακή Προεδρία και απέναντι στον Κυπριακό λαό. Δεν μπορεί να μας αποκαλούν ότι είμαστε φιλοί ή δεν είμαστε καν φιλοί. Αυτό το πράγμα δεν, περνε, δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητο. Πρέπει να επιρριφθούν ρητό ευθύνε για τη μη πραγματοποίηση τη 70 Συνόδου τη Μιχτής κοινοβουλευτική επιτροπή Τουρκία Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να επιρρευθούν ευθύνε για τι απειλέ εναντίον τη Κυπριακή Δημοκρατία για την προσπάθεια αξιοποίηση των ε, υποθαλασσίων ε, κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Και δεν μπορούμε να συζητάμε το άνοιγμα του κεφαλαίου για την ενέργεια όταν μα απειλούν ξεκάθαρα και δεν μα επιτρέπουν να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Τέλο, όσον αφορά το καθεστώ τη του, κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση παραμένει ω είχε και προηγουμένω. Καλείται μεν η Τουρκία να παραδώσει την πόλη στα Ηνωμένα Έθνη, καλείται παράλληλα και η Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι. Και αυτό είναι σωστό, γιατί μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να ανοίγει, τελειώνω πρόεδρε, να ανοίγει και να κλείνει τα λιμάνια και τα αεροδρόμια στη χώρα με ένα νομικό τρόπο, λέει, που να είναι αποδεκτό από όλε τι πλευρέ. Ο μόνο νομικό τρόπο είναι το διεθνέ δίκαιο είναι οι, οι δημοκρατικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η αντιδήλωση της 21 η ε, Σεπτεμβρίου δεν μπορεί να υπάρχει άλλο. Ευχαριστώ, θα ήθελα να πω περισσότερα, αλλά δυστυχώς πάντα είναι ασφιχτικό ο χρόνος για μα τους μικρούς. Ε, Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κινδυνεύω και εγώ να επαναλάβω όσα λέχθηκα. Αλλά ζούμε στην Κύπρο και βιώνουμε την κατοχή. Το θεμελιώδε δικαίωμα τη ελεύθερη διακίνηση, εγκατάσταση και εργασία σε ολόκληρη την επικράτεια τη Κύπρου παραβιάζεται από την κατοχική Τουρκία. Και φέτος είναι το 2013 Ευρωπαϊκό Έτο Πολιτών. Εγώ θα ήθελα μέσα στην έκθεση ακριβώ να μην υπάρχει αναφορά ότι και τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να κάνουν ε, τις δικές τους κινήσεις. Γιατί υπάρχει προσπάθεια, παρότι είναι πολύ καλή έκθεση, να υπάρχει ακριβώς ίση αντιμετώπιση και προς την κατοχική Τουρκία και προς το θύμα που είναι η Κύπρος. Και αυτό είναι λάθος. Προσωπικά θα κάνω κάποιες τροπολογίες, γιατί θέλω στην παράγραφο 24 να γίνεται αναφορά ότι δεν αρκεί μόνο να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια για το θέμα των αγνωμένων, πρέπει να πιεστεί η Τουρκία να ανοίξει στρατιωτικές ζώνες, γιατί καθημερινά ανοίγει νέες περιοχές που τις ονομάζει στρατιωτικές ζώνες για να μην μπορεί να γίνει ε, προσπάθεια για διακρύβωση της τύχης των αγνωμένων. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Θα ήθελα την κυρία Όμεν αυτήν την αναφορά για τις στρατιωτικές ζώνες, ζώνες να τη συμπεριλάβει. Επίσης, Όσον αφορά τη Σύνοδο, την 70η Σύνοδο, θεωρώ απαράδεκτο διότι ήταν μεγάλη πρόκληση να μην πραγματοποιηθεί, όχι εξυπαιτιότητα τη Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κυπριακή Προεδρία ήταν πολύ πετυχημένη. Προσπαθήσαμε να πάμε στην Τουρκία το δεύτερο εξάμεινο του 2012, δεν κατέστη εφικτό. Η Κυπριακή Προεδρία έκαμε προσπάθειες όσον αφορά την προώθηση ε, για τη βίζα των Τούρκων υπηκών και αυτό πρέπει να εκτιμηθεί, ενώ η Τουρκία απειλούσε την Κυπριακή ε, Προεδρία και για το θέμα της ΑΟΣ και για το φυσικό αέριο. Πρέπει να γίνει καταγραφή εδώ ποιο έφταξε. Γιατί τώρα σε λίγε μέρε, 11 με 15 του Φεβράρι, θα πάμε στην Τουρκία, λίγε μέρε πριν από τι προεδρικέ εκλογέ. Και δυστυχώ θα ακολουθήσουμε αυτό που λέγεται business as usual. Δεν είναι business as usual. Δεν μπορεί μια χώρα υπό ένταξη να παραγνωρίζει ευρωπαϊκού θεσμού. Θα μπορούσα να πω πολλά. Απλά θα πω ότι εκφιάζεται πολύ ο οικονομικός ρόλος της Τουρκίας. Να με επιτρέψετε όμως να πω ότι τα πολιτικά κριτήρια που είναι πολύ σημαντικά για την Ευρώπη των λαών και των αρχών παραβιάζονται. Θέμα καταπάτησης δικαιωμάτων των γυναικών, των δημοσιογράφων, καταγγελίες της διεθνούς αμνηστίας. Στη χώρα μου υπάρχουν σωρία τέτοιων παραβιάσεων. Επομένως, δεν συμφωνούμε με το άνοιγμα των κεφαλαίων και δεν γίνεται αναφορά μόνο για το το 23 και το 24. Στην έκθεση γίνεται αναφορά και για το άνοιγμα του 15 και του 22 και κάποιο ανάφερε και το 30. Λυπούμε να πω ότι με το να ανοίγουμε κεφάλαια και να θοπεύουμε την Τουρκία δεν θα λυθεί ποτέ το Κυπριακό. Thank you. Mrs. Gomes, Η κυρία Γκόμες. Πρώτα απ' όλα, η Τουρκία πρέπει να ενισχυθεί από εμά όσον αφορά την ανθρωπιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων στην περιοχή, τους πρόσφυγες κλπ. Συνεχίζονται οι συνομιλίες. Συμφωνώ πάντως ότι η δολοφονία των Κούρδων ε, γυναικών ε, στο Παρίσι είναι ένα μεγάλο χτύπημα. Χρειάζεται να ερευνηθεί το θέμα πλήρως και το δικό μας το κοινοβούλιο πρέπει να είναι σαφές ως προς αυτό. Πιστεύω ότι πράγματι και στηρίζω σε αυτό τη Ρία που πάντα μας προσφέρει πολύ ισορροπημένες ε, προσεγγίσεις και εκθέσεις όπως και τώρα Στηρίζω λοιπόν αυτό που λέει για το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24 και το να τεθούν στόχοι προς επίτευξη. Σίγουρα η Τουρκία μένει πολλά να κάνει. Έχουμε καταλήξει να έχουμε περισσότερους ε, φυλακισμένους ε, εκεί από ότι Κίνα, Ινδία. Είναι το πρόβλημα Ιράν. Είναι πολύ σημαντικό επίση να δούμε πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στη χώρα αυτή. Ο αντιτρομοκρατικό νόμος. Τώρα όμως θέλω να σχολιάσω το θέμα του Κυπριακού και να συγχαρώ την Κύπρο για τον τρόπο που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό κατά την Προεδρία της. Δηλαδή ότι κατάφερε να μείνει πιστή στους στόχους της χωρίς να βγει καθόλου από την πορεία της. Οπότε τώρα είναι απολύτως φυσιολογικό εμείς να πούμε στους φίλους μας στην Τουρκία ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοιου είδους συμπεριφορά και ότι μπορούμε να δεχτούμε τη θεωρία του business as usual πρέπει να τηρήσει το πρωτόκολλο. Και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκε κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας είναι απλώς απαράδεκτος για την Ευρώπη. Και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να εμποδίσουν την Κύπρο να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες για πετρέλαιο στο... στη θάλασσά της είναι επίσης κάτι το απαράδεκτο. Αυτό πρέπει να το πούμε και ελπίζω να συμφωνήσω και οι συνάδελφοι με μια πιο σκληρή γλώσσα. Συγχρόνως βέβαια πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε την ιδέα ότι τα κεφάλαια 23 και 24 πρέπει να ανοίξουν. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει αντίφαση από αυτού. Ευχαριστώ. Κρέσσελτορφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ και εγώ την συνάδελφο Όμεν Ρόιτεν για την συνεκτική, καλοδιατυπωμένη έκθεση. Προφανώς θα υπάρξουν και πολλές μάλιστα τροπολογίες, όσοι ήθιστε, ορισμένες βελτιωτικές σίγουρα. Χαίρομαι που βρίσκονται εδώ και οι φίλοι από την Τουρκία. Είναι καλό να αναδείξουμε μια κουλτούρα συζήτησης, διαλόγου, ε, που πάντοτε συμβάλλει θετικά στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υπάρχουν θέματα που τα επικρίνουμε όπως στην Λωρίδα της Γάζας, ε, στη Συρία. Εμείς όμως οι σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία τις διαπραγματεύσεις τις βλέπουμε προς την κατεύθυνση της προσχώρησης και όχι ε, μιας προνομιακής εταιρικής σχέσης ή οτιδήποτε άλλο ε, μπορεί να φανταστεί κανείς. Δεν είμαι κατά του ανοίγματο των κεφαλαίων 23 και 24 γιατί νομίζω ότι σε αυτούς τους τομείς η Τουρκία θα πρέπει να λύσει αυτά τα θέματα και για ίδιο συμφέρον, όχι μόνο για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καλό να βελτιωθεί το θέμα της, το θέμα της δικαιοσύνης, των εσωτερικών υποθέσεων, της ελευθεροτυπίας. Ε, αυτό το οφείλει η κυβέρνηση στον ίδιο της στο λαό. Παρ' όλα αυτά όμως καλό είναι να ε, συζητηθεί το ενδεχόμενο του ανοίγματο. Το Κυπριακό είναι βέβαια πολύ σημαντικό, αλλά θα πρέπει να συζητηθεί ε, με όριμο τρόπο. Εμείς ε, τώρα ε, έχουμε την, ε, φέτος την επέτειο της, του, της, του Γαλλογερμανικού Συμφώνου που ένωσε δύο κράτη τα οποία είχαν περάσει από πολλές διαιρέσεις και διχασμούς. Θα μπορούσε κάτι τέτοιο να επαναληφθεί. Ε, παρόλο που βεβαίως ε, και οι κλιματικές διαφορές ε, δημιουργούν διαφορές σε σχέση με τη σχέση των δύο χωρών ένθε και κήθεν. Ε, θέλω να συγχαρώ την κυρία Όουμεν, η οποία είναι ο επί των τουρκικών θεμάτων, ε, όντας εισηγήτρια επί πάρα πολλά χρόνια και παρακολουθώντας τα στενά. Πράγματι, η έκθεση είναι ισορροπημένη, αλλά δεν επαναλαμβάνει ορισμένα πράγματα για τα οποία η Τουρκία δεν συμμορφώνεται και δεν θέλει να συμμορφωθεί με κανένα τρόπο. Είναι τα ζητήματα της Άγκλος, της αποδοχής της συνθήκης του Μοντίγκο Μπέι, δηλαδή του δικαίου της θάλασσας, είναι τα ζητήματα που έχουν σχέση με τις απειλές περί πολέμου για την άσκηση δικαιωμάτων από την πλευρά άλλων χωρών, στην προκειμένη περίπτωση της Ελλάδος, και είναι μία σειρά ζητημάτων που αφορούν στις θρησκευτικέ ελευθερίες και στα δικαιώματα. Ε, πιστεύω ότι η κυρία Όμεν, ε, εγώ θα κάνω κάποιες λίγες τροπολογίες, πιστεύω ότι θα ενσωματώσει και αυτά, ίσως γιατί πρέπει να είναι χαρακτηριστικά κάθε χρόνο και να γίνεται αντιληπτό ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια αιμονή ε, σε θέματα βασικών δημοκρατικών αρχών, αφού μιλάμε για μια προοπτική ευρωπαϊκή και επίσης θα ήθελα μια διαφορετική διατύπωση στο άρθρο 3, στο σημείο ε, εκείνο ιδιαίτερα που υπάρχει το θέμα της επανεισδοχής, διότι κύριε Πρόεδρε, η συμφωνία που έχει γίνει περιλαμβάνει επανεισδοχή κατά τα τρία πρώτα έτη μόνο Τούρκων υπηκών και εν συνεχεία έπονται οι άλλοι και εκεί υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Δηλαδή απελευθέρωση, η πλήρης απελευθέρωση της βίζας στην Τουρκία ε, αν συνοδευτεί από αυτή την θέση που έχει τώρα η Τουρκία φοβούμε πως είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο χωρίς να πάρουμε ανταλλάγματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. Uh, Mr. Kachin, please. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κατσίν. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Όντως είναι ισορροπημένη η έκθεση, αλλά αυτό που πρέπει να προσθέσουμε εδώ είναι η αναγνώριση ότι πρέπει να εστιάσουμε στα θέματα που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Η Τουρκία πολλές φορές έδειξε ότι θέλει την πρόοδο ανάπτυξη και δημοκρατισμό και ελπίζω και νομίζω ότι θα βοηθήσουμε τον τουρκικό λαό ε, περισσότερο αν τους βοηθήσουμε να ανοίξουν τα απαιτητικά κεφάλαια. Χρειάζεται έλευθο βήμα να πέσει αυτός ο αποκλισμός, να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που έμειναν επί δεκαετίες και δεν μας βοήθησαν. Θέλουμε λύσεις τώρα. Ένα παράδειγμα, διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου-Πρίστινας. Η Σερβία δεν αναγνωρίζει το κοσυφοπέδιο, αλλά σε λίγους ε, μήνες μπόρεσε να κάνει ε, μεγάλο βήμα και τώρα άρχισαν άμεσες ε, συνομιλίες και η πρόοδος είναι καθημερινή. Αυτό ήταν αδιανόητο πριν από λίγους μήνες και όμως είναι μια σημερινή πραγματικότητα. Θα έπρεπε η Λευκοσία και η Άγγελα να κάνουν κάτι παρόμοιο και να καταρριφθεί αυτός ο αποκλεισμός. Η διαδικασία της διεύρυνσης του 2004 δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και αυτό είναι πρόκληση για όλους μας. Στο κάτω-κάτω η Τουρκία είναι σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, αλλά και στην, περιοχή γενικότερα. Ε, η τοποθέτηση πυράβλων πάτριων ε, είναι ένα δείγμα αλληλεγγύη μεταξύ Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει όμω να γίνουν συγκεκριμένα βήματα. Ε, πρωτίστως εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μάθουμε περισσότερα από την ικανότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεπέρασε την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση πριν από λίγα χρόνια. Είναι μεγάλη επιτυχία για τη χώρα και ως φιλελεύθερος υπογραμμίζω ιδιαίτερα την πρόοδο και την επιτυχία που πέτυχε, πέτυχε η Τουρκία στον εξυγχρονισμό ε, των γυναικών, τη συμπερίληψή του στην ε, εκπαίδευση, γιατί με τις γυναίκες στην παιδεία θα κάνει μεγάλο βήμα εκδημοκρατισμού, μετασχηματισμού και μεγάλου ανοίγματο. Η Τουρκία είναι ε, εκείνη που ε, βοηθεί την ευρωπαϊκή πολιτική στην περιοχή. Είναι ένας σύμμαχος και ένας φίλος μάλιστα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τέτοιος αν ε, είχαμε επιτρέψει ελεύθερη εκείνη στα Δυτικά Βαλκάνια και αν μπορούσαμε να έχουμε απελευθέρωση των θεωρήσεων εκεί, δεν βλέπω γιατί κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά στην Τουρκία η οποία χρειάζεται τη βοήθειά μας και εμείς πρέπει να επιδείξουμε περισσότερη τόλμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Χάουιτερ, καταρχήν χαιρετίζω το σχέδιο έκθεσης ε, η κυρία Όμεν Ρόιτεν προσπάθησε πραγματικά να δώσει μια βάση ισορροπημένη για να προχωρήσουμε εμείς περισσότερο. Ε, πολύ καλή είναι η αναφορά στην απελευθέρωση των θεωρήσεων στο 3. Επίσης πρέπει να υπάρξουν ορόσημα ή σημεία συγκριτικής αξιολόγησης και για το Κυπριακό συμφωνώ με τη συνάδελφο Άννα ε, που είπε ότι είναι πολύ καλή η Κυπριακή Προεδρία και Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει πειθαρχία, δεν θα πρέπει να είναι δυσανάλογη η έκθεση αυτή ε, στις αναφορές της Κύπρου. Ε, εις ό,τι αφορά την προσπάθεια βελτίωσης, ε, νομίζω ότι είχαν 10% ε, οικονομική ανάπτυξη, ε, τη μεγαλύτερη στην περιοχή. Συμφωνώ και επίσης σε σχέση με τον κεντρικό ρόλο της Τουρκίας ε, σε σχέση με την Συρία και τους ε, πρόσφυγες από εκεί. Ίσως αυτό πρέπει να το αναδείξουμε περισσότερο. Για το διαμεσολαβητή νομίζω ότι δεν ε, επικρίνει τον περιορισμό των εξουσιών του διαμεσολαβητή, έρευνες σε σχέση με τις φυλακές που και μάλιστα σε μια ψηφοφορία το κόμμα της αντιπολίτευσης, το CHP, δεν συμμετείχε και ε, το θέμα το χειρίστηκε μόνο το κυβερνητικό κόμμα. Ε, Επίση σε σχέση με το κουρδικό, ε, εγώ είχα παρακολουθήσει δίκες του CKC και νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην χαθεί η ευκαιρία που ανοίγεται τώρα στο Κυπριακό. Τώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα η αντιπροσωπεία στην Άγκυρα προσπάθησε να ε, ακολουθήσει κοινέ κατευθυντήριες γραμμές. 18 Ιανουαρίου φέτος ε, επίσης ε, διώχθησαν ε, αρκετοί δικηγόροι και αυτό είναι πλήγμα για μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Λάντφορντ. Ζητώ συγγνώμη που άργησα και δεν άκουσα την εισηγήτρια και τους περισσότερους Όδησε. Νομίζω ότι είναι καλό σχέδιο έκθεσης, ισορροπημένο, ε, αρκετά συνεκτικό, σύντομο, όλα αυτά είναι θετικά. Συμφωνώ με την αναγκόμες των Ρίτσορ Χάουιτ που είπαν ότι θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο κάποια θετικά στοιχεία ε, δηλαδή θέματα οικονομικά, ανάπτυξη, θέματα εμπορίου, ο θετικός ρόλος της Τουρκίας νομίζω ότι ε, ίσως θα έπρεπε στην ε, ε, δεύτερη σελίδα να επικεντρωθούμε σε αυτά. Βεβαίως δεν θα υποβαθμίσουμε, δεν θα περιορίσουμε την κριτική μας, αλλά τα θετικά να γίνουν πιο ορατά. Επίσης, στην παράγραφο 9 που γίνεται αναφορά στις απειλές κατά της ελευθερίας έκφρασης, της σύλληψης των δημοσιογράφων, εδώ το θέμα είναι πραγματικά πολύ δύσκολο και έχει αναφορές στο κουρδικό. στο οποίο πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Να Ε, υπάρξει ε, υποστήριξη για ε, εξέβρεση πολιτικής λύσης. Πρέπει να αναφερθούν βέβαια και οι δολοφονίες στο Παρίσι, αλλά και συλλήψεις που γίνονται σε κάποια κράτη-μέλη της Ένωσης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η δίωξη της τρομοκρατίας του ΠΚΚ δεν θα υπονομεύει τις πολιτικές δραστηριότητες των Κούρδων ακτιβιστών υπέρ της αυτοδιάθεσης και αυτονομίας. Τέλειωσε ο χρόνος. Τέλειωσε. Δύο λεπτά δεν είχα. Α, δέκα δεύτερα λεπτά. Ε, για την απελευθέρωση των θεωρήσεων ε, ήθελα επίσης να πω αλλά αναφέρθηκε και από άλλους. Τώρα, για την Κύπρο, συμφωνώ με κάποιες παρατηρήσεις που ακούσαμε, αλλά είναι ατύχημα το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία κάνει ε, προσπάθεια, ε, ε, έχει PDO για το χαλούμι και να αποκλείσει το χαλίμ που είναι το ίδιο τυρί το οποίο ε, παρασκευάζεται ε, στη Τουρκία. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν περισσότερο στο ζήτημα αυτό με το τυρί. πρόεδρος της ε, Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ευχαριστώ, λέει κυρία Φλότρο. Άργησα εξαιτία του χιονιού. Γι' αυτό και Λείπουν κι άλλοι βέβαια. Λοιπόν, για να επανέλθω στη συζήτηση για την Τουρκία. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ την κυρία Όμεν Ράιτεν. Είναι συνέχεια στη δουλειά που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια για να ενισχύσουμε τη συνένεση την οποία έχουμε αρχίσει να πετυχαίνουμε ήδη από τις προηγούμενες εκθέσεις και προχωράμε και τώρα και μιλάμε για άνοιγμα νέων κεφαλαίων, κάτι το οποίο είναι όχι μόνο επιθυμητό αλλά και εφικτό. Σήμερα είμαστε μπροστά σε ένα πολιτικό παράθυρο έξι μηνών και νομίζω ότι αυτή πρέπει να τη δούμε, αυτό το άνοιγμα πρέπει να το δούμε σαν μια πραγματικά μεγάλη πολιτική ευκαιρία για να προχωρήσει η διαδικασία ένταξη τη Τουρκία και να ενισχυθούν οι σχέσει τη Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και πρέπει να υπογραμμίζουμε στην έκθεση αυτή τα διάφορα ευαίσθητα σημεία, το κουρδικό για παράδειγμα, το θέμα των ε, μεταρρυθμίσεων στο τομέα της δικαιοσύνης, ε, να λέμε για την σημασία που δίνουμε στην εκπόνηση του νέου συντάγματος, στην ελευθερία έκφραση των δημοσιογράφων και υπάρχουν κάποια σημεία στο οποίο μπορούμε να βαθύνουμε ακόμα περισσότερο το κουρδικό, όπως είπα και πριν. Υπάρχει κάποια διαδικασία, είναι καλό που υπάρχει να την ενθαρρύνουμε και να μην ε, μπαίνουν εμπόδια όπως οι πράξεις αυτές στο Παρίσι, δολοφονίες στο Παρίσι. Υπάρχει τώρα το θέμα της ενίσχυσης των δικαιωμάτων. Ελπίζουμε ότι θα προβλέπονται στο νέο σύνταγμα βέβαια. Η ελευθερία έκφρασης ε, και η γνώση της μητρικής τα αξιώματα που θα μπορούν να κατέχουν στην κοινωνία. Αλλά πρέπει να δούμε και το θέμα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και τον πολιτικό διάλογο προς αυτή την κατεύθυνση. Το διάβασα βέβαια, θα το κρίνει από μόνη της η κυρία Όμεν Ράτεν. λοιπόν διαβάζοντας το κείμενο μήπως μπορούμε να βαθύνουμε περισσότερο τα περί ελευθερίας του τύπου και ελεύθερη έκφραση. Μήπως να μιλήσουμε για την ε, Επιτροπή ΑΤΟΚ που είχαμε για αυτό το θέμα, γιατί έχει γίνει αρκετή δουλειά από τους ευρωβουλευτές πάνω σε αυτό. Πολλές αναλύσεις. Ίσως λοιπόν μπορούμε να το αναφέρουμε στην έκθεση. Ευχαριστώ κατά τα άλλα την κυρία και μπορεί να βασιστεί σε μένα για να στηρίξω τη γραμμή που επέλεξε, που είναι μια γραμμή ανοίγματο, ανοίγματο συζητήσεων για το κουρδικό, ανοίγματο νέων κεφαλαίων και γενικά άνοιγμα προς την κατεύθυνση του νέου συντάγματος. Αυτή είναι πράγματι η γραμμή που πρέπει να ακολουθήσουμε σήμερα, πιστεύω. Είναι σωστή και θα είναι και καρποφόρα. Γιατί βέβαια θέματα όπως είναι το κουρδικό είναι θέματα που τίθενται γενικότερα στην περιοχή και στη Συρία και στο Ιράκ, άρα είναι γεωπολιτικό το θέμα και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό στην έκθεση αυτή να τονίζουμε την πολιτική μας δέσμευση ώστε να συνεισφέρουμε σε μια, με αποφασιστικό τρόπο σε μια λύση. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης για την Διεύρυνση τώρα. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ε, Ευχαριστώ πολύ και σας και την εισηγήτρια. Θέλω να χαιρετήσω εδώ πρώτα απ' όλα το έργο της Omen Writer. Έχει ετοιμάσει μια ισορροπημένη έκθεση, μια σωστή έκθεση και από πλευράς ουσίας αλλά και από πλευράς ύφους. Η έκθεση αυτή αντιστοιχεί απόλυτα στα συμπεράσματα της έκθεσης πρόοδου που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2012 και αντικατοπτρίζει επίσης και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που υιοθετήθηκαν τον Δεκέμβριο. Η θετική ατζέντα πιστεύουμε ότι έπαιξε έναν αποφασιστική σημασία ρόλο για να διατηρηθούν οι σχέσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία στο σωστό δρόμο. Παρά τα διάφορα προβλήματα, τις διάφορες ε, δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε τον τελευταίο καιρό και στις οποίες αναφέρθηκαν οι προλαλήσαντες. Μόνο να αναφέρω το ότι ολοκληρώθηκε ο χάρτης πορείας όσον αφορά την ελευθέρωση του καθεστώτος ε, θεωρήσεων για τους Τούρκους υπηκόους. Όλα αυτά ε, συνσέφεραν και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου που λέει ότι πρέπει να κοιτάμε προς το μέλλον. Επικοδομητικά λοιπόν συμπεράσματα τα οποία ετοιμάζουν το δρόμο για μια νέα όθηση των συνομιλιών εν ώψη της ένταξης της ε, Τουρκίας. Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι πήραν το λόγο εδώ για να μιλήσουν υπέρ των ανοίγματο των κεφαλαίων 23 και 24. Εμείς πιστεύουμε ότι μόνο ανοίγοντα τα κεφάλαια αυτά μπορούμε πραγματικά να έχουμε ένα διάλογο πιο εντατικό με την Τουρκία για να διακανονιστούν όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα ή με την δικαιοσύνη, ό,τι άλλο αναφέρατε εσείς σχετικά. Όλα τα θετικά που αναφέρει η έκθεση της κυρίας Όμεν Ράιτεν που ενθαρρύνουν τη χώρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση πιστεύουμε εμείς και θέλουμε να ενθαρρύνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης στην Τουρκία για την πρωτοβουλία της προκειμένου να τελειώσει αυτή η αιματηρή περίοδος όλες αυτές τις δεκαετίες και να υπάρξει μια συνολική λύση για το κουρδικό. Γιατί έτσι θα λυθούν και άλλα πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα πολιτικά κριτήρια τα οποία έχουμε στις εκθέσεις μας και συζητάμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Πριν ζητήσω από την εισηγήτρια, την κυρία Ρία Όμεν Ράιτον, να κλείσει τη συζήτηση, θέλω να σας υπενθυμίσω προθεσμία για την, για την ε, προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι η 5η Φεβρουαρίου 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μαζί με τους συνεργάτες μου προσπάθησα να παρουσιάσω μια ισορροπημένη έκθεση για την πρόοδο της Τουρκίας. Ισορροπημένη αλλά επίσης ειλικρινής παρατηρήσεις. Η έκθεση, θα ήθελα να πω σε όλους, είναι αποδεκτή από την μεγαλύτερη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, μεγάλη πλειοψηφία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. 90% ήδη είχαμε, που είχαμε μάλλον ανέκαθεν και ελπίζω πως και αυτή τη φορά το ίδιο ποσοστό θα επιτύχουμε. Ε, δεύτερη μου παρατήρηση είναι πως θα ήθελα να θυμίσω άλλη μια φορά εδώ πως οι διαπραγματεύσεις είναι ανοιχτές. Και δεν μπορούμε τώρα να δώσουμε ημερομηνία. Καταρχήν ε, τα πολιτικά κρατητήρια θα πρέπει να πληρώνται. Διότι αυτό είναι το βασικότερο θέμα. Είναι ακόμα πιο σημαντικό από την συζήτηση των κεφαλαίων. Για να στραφούμε στα κεφάλαια. Εάν θέλουμε η Τουρκία να κάνει περισσότερα για το δικαστικό σώμα, να κάνει περισσότερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε θα ήταν καλό, είναι καλό να έχουμε θετική ατζέντα και να έχουμε κάποιες άτυπες ε, άτυπου πίνακε ε, επιδόσεων και γι' αυτό χρειάζεται το άνοιγμα αυτών των κεφαλαίων. Τρίτον, ελεύθερο, ελευθερία των μαζικών μέσων ενημέρωσης και έκφρασης. Είναι βασικές ευρωπαϊκές αξίες θα έλεγα. Και γι' αυτό τονίζουμε στο άρθρο 9 ότι χρειάζεται μια, οπωσδήποτε μια μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα το τέταρτο πακέτο και ό,τι έχω δει θα μπορούσαν να μας φέρουν σε κάτι τέτοιο. Επίσης πριν από μια μισή εβδομάδα είχα συζητήσει με το Συνταγματικό Συμβούλιο, με το, είπα, το Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων και επίσης με τον Σύνδεσμο Δικαστών και είμαι πεπισμένη πως η Τουρκία θέλει κάτι να κάνει. Ενέργεια. Εάν η Τουρκία μπλοκάρει τη συμμετοχή της Κύπρου και του Ισραήλ στον Οργανισμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι χώρες αυτές θα πρέπει να θυμηθούν ότι, ότι τα κεφάλαια ενέργειας είναι μπλοκαρισμένα από τις ίδιες. Ε, θα πρέπει λοιπόν να απεμπλακούν και ελπίζω πως η πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο θα υπάρξει. Ναι, τώρα για ε, τον ΟΑΣΕ και τον Ιδωμένο για ε, τη Συμφωνία για τη Θάλασσα των Εθνών θα το, θα το αναφέρω σε μια παράγραφο. Τώρα, άμεσα τι θα πρέπει να γίνει. Στη Τουρκία και τα αυτά τα πρωτόκολλα θα επικυρωθούν, αλλά θα μπορούσες και να διαρωτηθείς εσύ, Τσάλς, γιατί δεν έχουν επικυρωθεί. Λόγω των κακών σχέσεων γυτνίασης με κάποιες χώρες. Ας κάνουμε λοιπόν κάτι για να ξεμπλοκάρουμε την κατάσταση, γιατί για μένα η προτεραιότητα είναι το άνοιγμα των συνόρων. Ε, τώρα, για το περιβάλλον και την οικολογία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ με... βασικά μίλησα για κάποιους χαρακτήρες, αλλά εάν υπάρχουν ε, ε, με δέσμευαν μάλλον οι χαρακτήρες στην έκθεση για το μάκρος έκθεσης, αλλά αν υπάρξουν τροπολογίες θα τις λάβω υπόψη ε, τα κεφάλαια τα 23 ε, και 24 για το κράτος δικαίου συζητούνται στο τέλος της διαδικασίας για το κουρδικό ζήτημα. Νομίζω πως ήμουν αρκετά σαφής πως η ε, δολοφονία στο Παρίσι ήταν μια απλή πρόκληση. Απλή πρόκληση, ξεκάθαρη πρόκληση για την ε, πολιτική διαπραγματευτική διαδικασία ανάμεσα στην τουρκική κυβέρνηση, τους εκπροσώπους της τουρκικής κυβέρνησης και του κύριου Οτσαλάν. Ήταν μια ξεκάθαρη πρόσκληση και πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να γίνει μια καλή έρευνα. Ε, αλλά δεν είναι αυτό όλο. Η έρευνα πρέπει να γίνει στο Παρίσι. Και από ό,τι άκουσα, δεν ξέρω αν είναι φήμη ή όχι, έχει ήδη γίνει μια σύλληψη σήμερα. Κάποιου που προέρχεται από το ΠΚΚ. Τι να πούμε παραπάνω. Εγώ δεν θέλω να διαταραχτεί η διαδικασία ειρήνης στην Τουρκία και γι' αυτό τον λόγο νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είμαστε βέβαια να μην σιωπήσουμε αλλά να προσέξουμε πάρα πολύ τι θα πούμε. με Κοπά. Είμαι κάθετα αντίθετη στο ότι η Τουρκία δεν δέχτηκε την Κύπρο ως αρχηγό στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Τι να κάνω άλλο. Ήμουν κάθετα αντίθετη, όχι μόνο γραπτός στο κείμενο, αλλά και όταν μίλησα για το θέμα αυτό. Τέλος, για το θέμα Τουρκία-Συρία. Εγώ επισκέφθηκα δύο στρατόπεδα προσφύγων και το συζήτησα με τον επίτροπο που είναι υπεύθυνο. Και, και εκείνη, ή που είναι υπεύθυνη, ε, και εκείνη συνεχάρει την Τουρκία για τον τρόπο με τον οποίο οργάνωσε τα πράγματα. Γιατί η κατάσταση που είδα εγώ σε αυτά τα δυο στρατόπεδα προσφύγων ήταν καλύτερη από ότι αλλού. Αγνοούμενοι. Αγνοούμενοι, όχι, δεν, ε, τους ανέφεραμε, ναι. Για τον διαμεσολαβητή. Ήξερα, γνωρίζω μάλλον, ότι υπάρχουν κάποια σχόλια όχι μόνο για τις αρμοδιότητες αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο διορισμός. Αλλά αυτό που εγώ θέλω να δω είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Οπότε ας την κρίνουμε τον επόμενο χρόνο. Προσπάθησα, όπως είπα, να κρατήσω ισορροπία στην έκθεση και αν έρχεται ο καθής με μια μονόπλευρη τροπολογία, θα κάνω ό,τι μπορώ να διατηρήσω αυτή την ισορροπία. Αν έχει γίνει καλή την πίστη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Μενρό. Ήταν ευχαριστώ συνάδελφοι. Ας μην ξεχνάμε ότι αύριο αρχίζουμε στις 9 με τις ψηφοφορίες. Τέλος της συνεδρίασης. Nine.